Se prendete posto, per favore, cominciamo. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ πολύ προκειμένου να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Non comincio. Io comincio, mi importa. Allora, buongiorno a tutti, se vi accomodate per favore cominciamo. Grazie. Καλημέρα σας και πάλι. Καθίστε παρακαλώ πολύ ώστε να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Il progetto di ordine del giorno di questo incontro Έχουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης για τη σημερινή συνεδρίαση, το οποίο σας απεστάλλει στις 20 Οκτωβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γνωρίζετε επίσης ποιο είναι το γλωσσικό καθεστώς. Η συνεδρίαση επίσης ε, πρόκειται να μεταδοθεί ζωντανά. Μου είπαν χθε το βράδυ ότι ο πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, κύριο Καλτέρα, θα φτάσει λίγο αργότερα από ό,τι προβλέπετε. Μετά από αίτημα του κυρίου Μπούζεκ που θα τον υποδεχθεί στι 9.30 αντί στι 9 προβλεπόταν αρχικά. Μα ζητήθηκε λοιπόν να περιμένουμε λίγο παραπάνω τον κύριο Καλτέρα, τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης παρουσίαση των οριστικών νοποιημένων ετήσιων λογαριασμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008. Ο κύριος Φιλίπ Ταβέρνη είναι ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του δίνω κατευθείαν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ο προκάτοχο μου ο κύριος Γκρέ ανέλαβε την θέση του υπολόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και εγώ εξ ονοματός του θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω τους αριστικούς συνοποιημένους αιτήσεις λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008. Θα γνωρίζετε ότι πρόκειται να παρουσιάσουμε τον ισολογισμό, καθώς επίσης και το δημοσιονομικό δελτίο, το οποίο θα παρέχει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης και μια συνολική παρουσίαση των εσόδων και των δαπάνων, δαπανών για το έτος 2008. Παρουσιάστηκαν οι οικονομικοί αυτοί λογαριασμοί και καταρτίστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν το 2005. Βλέπουμε ότι το λογιστικό αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και λαμβάνει υπόψη του μόνο τις εκταμιεύσεις και τις πληρωμές. Οι ενοποιημένοι αυτοί οι λογαριασμοί για το 2008 αφαιρούν 39 ενότητες, τρία joint ventures και μία συνδεδεμένη οντότητα και έχουμε τρεις επιπλέον υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτήν για τις χημικές ουσίες, την υπηρεσία για την ενέργεια καθώς επίσης και την υπηρεσία για τις μεταφορές που είναι εκτελεστική υπηρεσία με την θέση σε ισχύ της θήκης της λαδώνας θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο νοποημένων λογαριασμών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή της άμυνας, του Κέντρου Δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας. Ποια, είναι η βασική, τα βασικά αριθμητικά στοιχεία. Βρισκόμαστε σε πλεον, πλεόνασμα του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, πράγμα το οποίο οφείλεται σε εκτέλεση κάποιων δαπανών σε κάποιους τομείς, όπως για παράδειγμα στα διορθωτικά ταμεία, στη γεωργική πολιτική, αλλά και στον τομέα της έρευνας. Το οικονομικό αποτέλεσμα φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ και πάλι εδώ πέρα μολονότι ακολουθήσαμε διαφορετικούς κανόνες κατάρτισης οι βασικέ αλλαγέ που έχουμε εδώ πέρα έχουν να κάνουν με μια σημαντική μείωση των δαπανών όσον αφορά τι διαρθρωτικέ δαπάνε με το τέλο των προγραμμάτων 2000-2006, ενώ υπήρξε μικρότερη πρόοδο από ό,τι προβλεπόταν για το πρόγραμμα 2007 2013. Έχουμε μείωση κατά 47 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το, τα θετικά του ισολογισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και έχουμε μία αύξηση της προχρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και τη γεωργική ανάπτυξη. Τέλος, όσον αφορά τα δάνεια τα οποία δόθηκαν και τα δάνεια τα οποία λήφθησαν, εδώ πέρα έχουμε ένα ποσό που φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο αντικατοπτρίζεται στον ενωπημένο ισολογισμό. Το 2008 είδαμε μια πολύ σημαντική αύξηση της προχρηματοδότησης, μια μείωση των βραχυπρόθεσμων ποσών και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μικρότερες δαπάνες οι οποίες αναλήφθησαν. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να αναφερθώ σε τρία βασικά ερωτήματα τα οποία τέθησαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το τα αρνητικά θετικά στοιχεία του προπολογισμού, τα αρνητικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και η απαραίτητη χρηματοδότηση όσον αφορά τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, βάσει των βασικών προδιαγραφών λογιστικών εκθέσεων, εργαζόμαστε βάσει ενός ετήσι, μιας ετήσιας έκθεσης προπολογισμού. Τα λογιστικά πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται ύψας FRS και πιο συγκεκριμένα οι κανόνες 3, 5 και 12 προβλέπουν συγκεκριμένη κατάρτιση του προπολογισμού που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στο τέλο του έτου όλε τι δαπάνε που σχετίζονται με το έτο αυτό, καθώ επίση και όλα τα χρέη και τα δάνεια τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες ΦΕΑΓΑ, καθώς επίσης και οι δαπάνες προσωπικού, χρηματοδοτούνται μόνο από το μελλοντικό προπολογισμό, από τη στιγμή που δεν εμφανίζονται στον τρέχοντα προπολογισμό. Οι ίδιοι λογιστικοί κανόνες δεν μας επιτρέπουν να συμπεριλάβουμε τις, τα μελλοντικά έσοδα ως χρέη στον υφιστάμενο προπολογισμό. Έτσι λοιπόν το σύνολο του παθητικού ξεπερνά το ενεργητικό και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα καθαρό ενεργητικό θετικό, το οποίο θα είναι αρνητικό, με συγχωρείτε. Όσον αφορά το 2008, το πρόγραμμα Γαλιλαίο δεν περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή γιατί βρίσκεται ακόμα σε φάση εξέλιξης, διαμόρφωσης και δεν μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να αντικατατροπηθεί δημοσιονομικά στον τρέχοντα προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται πολύ στενά με την ειδική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το πρόγραμμα Γαλιλαίο, προκειμένου τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος αυτού μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό και Βάσει τη μεταφορά αυτή θα καταρτιστεί μια έκθεση που θα μα επιτρέψει να αξιολογήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματο αυτού. Όσον αφορά την ε, απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή κτηρίων και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων για την κατασκευή αυτή. Ακολουθούμε πάλι δημοσιονομικού κανόνε που προβλέπουν ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο προπολογισμό παρά μόνο αν υπάρξει μια νομική απόφαση πριν την ολοκλήρωση του υποκατάρτιση προπολογισμού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η μελλοντική χρηματοδότηση για τα κτίρια αυτά και για τη συντήρηση των κτιρίων δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ενταχθεί στον υποεξέταση προπολογισμό. Για τα σημεία λοιπόν αυτά η λογιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά το οικονομικό καθεστώς Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης, χρησιμοποιώντας τους διεθνείς κανόνες ε, λογιστικής κατάρτισης. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολουθούσε τους κανόνες αυτούς, θα λάμβανε πολύ αυστηρή κριτική. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, μετά την εξέταση της αξιοπιστίας των ε, λογαριασμών αυτών, όλοι οι απαραίτητε πληροφορίες για την κατάρτιση των λογαριασμών, τόσο για το τμήμα του ενεργητικού όσο και για το θύμα και το τμήμα του παθητικού και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι ε, οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν μια πιστή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις σημαντικές πτυχές τους. Οι ονειπημένοι ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό του 2008 εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον ε, άρθρο 128 και 129 του Δημοσιονομικού Κανονισμού απαιτείται σημαντικό χρόνο καθώ επίση και προσπάθειε και προσαρμογέ προκειμένου να περάσουμε από ένα προπολογισμό στην πραγματική εκτέλεση του προπολογισμού αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει τι απαραίτητε προσπάθειε τον τελευταίο καιρό προκειμένου να βελτιώσει τη μετάβαση αυτή. Ιδίω λαμβάνοντα υπόψη κάποιε απόψει του ελεκτικού συνεδρίου στο παρελθόν που είχαν εντοπίσει ή μη σωστή εκτέλεση του κοινωνικού προπολογισμού. Σαφώ λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη τι συστάσει αυτέ του ελεκτικού συνεδρίου και είμαστε σε συνεχή επαφή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τι υπόλοιπε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιώσουμε τη χρησιμοποίηση των αιτήσεων αυτών λογαριασμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο το οποίο μα επέτρεψε να βελτιώσουμε την ποιότητα της οικονομικής μας κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δίνει την απαραίτητη προσοχή στις μελλοντικέ συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Επίτροπος κ. Κάλλας είναι εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράσκη. Θα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα καταρχήν να παρακαλέσω να παρακαλέσω να μπορέσω να δηλώσω πρώτα ότι η έκθεσή μου δεν πρόκειται να είναι πλήρης και διεξοδική διότι την Παρασκευή το απόγευμα βρισκόμουν στη Βασοβία ακόμα και το αεροπλάνο μου στις 9.30 το βράδυ ε, αναχώρησε. Το κείμενο μόνο το μεσημέρι το έλαβα. Το μεσημέρι όταν είχα φτάσει ήδη στις Βρυξέλλες αυτό το κείμενο μπόρεσα να το εξετάσω με μια πρώτη ματιά. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ την κατανόησή σας. Γι' αυτό η τοποθέτησή μου θα είναι πολύ σύντομη. Θα τοποθετηθώ πολύ σύντομα όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο. Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο και ακριβέστερες μελέτες. Πρώτα απ' όλα κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα λοιπόν, πρόοδος. Πρόοδος όσον αφορά την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχία. Ο αγωγητής διακόπτεται. Κάνουμε λόγο για το σημείο 3, εντάξει. Πρόκειται όχι για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, εντάξει ναι, εντάξει, λοιπόν, σύμφωνοι. Πράγματι, υπάρχει πρόοδος, λοιπόν, πρέπει να πω. Πρόοδος όσον αφορά την δημοσιονομική πειθαρχία, συνολικά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή όσον αφορά την διαχείριση του προϋπολογισμού από πλευράς διοίκησης και τα, την αντιμετώπιση των κονδυλίων έχουμε βελτιώσεις αλλά επίσης βελτιώσεις όσον αφορά και το σχέδιο του προϋπολογισμού και την εκτέλεσή του, την εφαρμογή. Προσεγγίζει το ένα σκέλος το άλλο. Ο κύριος ε, Διευθυντής έκανε λόγο για πέντε τομείς, για πέντε κλάδους. Φυσικά τι συμβαίνει εδώ αυτή μέσα στην παγιωμένη έκθεση του, πάγια έκθεση του 2008 εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποια προβλήματα και τριβές. Πρώτον, το ποσοστό σφάλματος. Και φυσικά στη συνέχεια έχουμε και αυτό το οποίο ίσως αφορά τον έλεγχο τον έλεγχο για την σωστή εκτέλεση δαπανών. Έτσι θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε το θέμα αυτό. Διαθωτικά ταμεία, διαθωτικά ταμεία, περιφερειακή πολιτική, πολιτική συνοχής. Είναι τομεί αυτοί όπου 200 έχουμε προβλήματα και 200 υφίστανται τριβές. Είναι προβληματικά πεδία αυτά. Πρώτον, το ποσοστό σφάλματος. Στη συνέχεια τα μέσα τα οποία στις προηγούμενες εκθέσεις ε, θεωρήθηκε ότι δαπανήθηκαν αχρέωστα και ε, αδικαιολόγητα και ε, κατανοώ βέβαια πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι οι δυσχέρειες αυτές έγκυνται στο ότι οι κυβερνήσεις συχνά το σύνολο αυτό το θεωρούν σαν μια ροή κονδυλίων, δημοσιονομικών κονδυλίων σε περίοδους κρίσης φυσικά σε κύρια ε, ε, έτη που πλήττονται από την κρίση έχουμε ε, το πρόβλημα όσον αφορά τα κονδύλια και Φυσικά έχουμε και την ισχύ, την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έναντι πολλές φορές των κρατών μελών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική και γνωρίζουμε εδώ ότι σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις και έτσι λοιπόν θα έλεγα μετά από τις τοποθετήσεις του κυρίου Αντιπροέδρου Κάλλας θα έλεγα θα έπρεπε να ε, δώσουμε σαφώς υποστήριξη εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να αξιολογήσουμε και να δούμε πόσο σημαντική είναι η εδραίωση των πραγμάτων, με παγιωμένη αντιμετω... πάγια αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι εξίσου σημαντικό αυτό όπως τα πρόσθετα κονδύλια, τα, τα πρόσθετα κονδύλια τα οποία ζητείτε να επιστραφούν, να ανακτηθούν. Και πόρο απέχουμε ακόμα από τις ιδανικές λύσεις δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τα, ε, την εκτέλεση. Είναι σαφές όμως ότι είναι σαφώς χαμηλότερο το ποσοστό σφάλματος από ότι σε σχέση με το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθεί να υφίσταται αυτό σε υψηλό θα έλεγα σχετικά επίπεδο και έτσι δεν είναι σαφές το τι ακριβώς συμβαίνει πάντα πρέπει να αποσαφινιστούν πολλά πράγματα. Εξάλλου έχει προγραμματίσει συγκεκριμένα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να δημιουργούν κινδύνους για την έρευνα. Σαφείς πρόοδοι έχουν σημειωθεί. Όμως έχουμε επίσης και το αρνητικό όσον αφορά το καθαρό ε, ε, ποσό των νεκρών. Αυτό αφορά τις ε, δαπάνες έρευνα. Θα ήθελα να πω λοιπόν έχουμε και ταμεία όπως ε, το Ajax, το Ajax που αφορούν για παράδειγμα την ε, Γεωργία. Υπάρχει σαφής βελτίωση που σημειώνεται. Σαν συνέπεια όλων αυτών θα ήθελα να παρακαλέσω το εξή. Κυρίε και κύριοι, αυτέ οι παρατηρήσει είναι πρώτε, ε, θα έλεγα, παρατηρήσει σε μια πρώτη φάση. Δεν μπόρεσα να προετοιμάσω τίποτα περισσότερο σε σχέση με το έγγραφο που πολύ πρόσφατα πήρα στα χέρια μου και πρέπει να ακούσουμε και τις, επι... Ε, τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για αυτή την έκθεση και θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις, κυρίως όσον αφορά το θέμα της ανάκτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Έχουμε το πρόβλημα ότι σύμφωνα με τα όσα γίνονται για την ανάκτηση είναι πολλές φορές αντιφατικά. Και αν δει κανεί ε, μετά από το ε, σχετικό εδάφιο το όσα αναφέρονται, έχουμε αυτό το πρόβλημα των αριθμητικών, των αριθμών, των ποσών. Θέλουμε σε σχέση με τις διαφορε... διαφορές μεταξύ γενικών διευθύνσεων να επιλύσουμε τα προβλήματα. Αυτό θελήσαμε να κάνουμε το παρελθόν, κατά το παρελθόν. Ήταν πρόθυμο και το ελεκτικό συνέδριο. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσον έχουν οριμάσει αυτές οι προσπάθειες. Πότε μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα έχουμε αξιόπιστα ποσά τα οποία θα υποβάλλονται χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Και αναφέρεται και στην αντίστοιχη σελίδα ότι ο κίνδυνος διαφορετικών αριθμητικών μεγεθών και ποσών υφίσταται. Πότε θα έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με τα ανακτώμενα ποσά, αξιόπιστα ποσά ε, στα οποία θα μπορούμε να βασιστούμε. Η πρώτη μου ερώτηση αυτή. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το σύνολο, το άθροισμα το οποίο θα πρέπει να ανακτηθεί. Εδώ γρήγορα, εντάχει είδα αυτό. Τι θα έπρεπε πάλι να γίνει ώστε στα επιμέρους ταμεία να γίνει για την ανάκτηση και ποιο θα είναι το ποσοστό συνολικά. Γνωρίζουμε ότι από άλλε πηγέ, για παράδειγμα από άλλε υπηρεσίε καταπολέμηση απατών, την Όλαφ, ότι στα αγροτικά, στις αγροτικές δαπάνες 20% από τα ανακτώμενα τελικά ανακτώνται. Δηλαδή, όποιος παίρνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη βεβαιότητα σχεδόν ότι θα μπορεί να τα διατηρήσει αυτά τα κονδύλια. Αυτό δεν είναι απόλυτα αποδεκτό, δεν είναι απαράδεκτο. Τι γίνεται σε εσείς με το σύνολο των ανακτώμενων ποσών. Θα ήμουν ευτυχή αν μα δίνατε αυτά τα αριθμητικά μεγέθη, αυτά τα ποσά. Ποιο είναι το ποσοστό των ανακτώμενων από τα επιμέρου ταμεία των επιστρεφόμενων κονδυλίων. Και για τα διαθροτικά ταμεία, εδώ δύο στοιχεία δεν μπορώ να τα καταστήσω συμβατά. Το, τα, τα 3,3 δις ευρώ εκεί κάτω στην αντίστοιχη σελίδα που πρέπει να ανακτηθούν λέει και το 1,58 δις ευρώ στη σελίδα 107 κάτω-κάτω. Ίσως θα μπορούσε κανείς αυτή την αριθμητική διαφορά αριθμητικών μεγεθών 1,1 δις για την ίδια περίοδο πώς μπορεί να εξηγηθεί το ότι υφίστανται διαφορετικά ποσά όσον αφορά την περίοδο ε, μέχρι το 2006. Ευχαριστώ. Grazie. Onorevole σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Ταβέν για την εξαιρετικά ακριβή παρουσίασή του και Εξάλλου, για το σύνολο των ε, προσαρτημένων σημειωμάτων ε, στους ε, παγιωμένους λογαριασμούς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Καταρχήν για τη μορφή. Οι αιτήσεις λογαριασμοί δεν έχουν μεταφραστεί. Θα ήταν δυνατόν να έχουμε τουλάχιστον σε κάποιες γλώσσες τη μετάφραση του εγγράφου, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε περισσότερο τόσο οι ευρωβουλευτές όσο και οι πολίτες. Επίσης, επί του τύπου με εντυπωσιάζει εξαιρετικά αργή διαδικασία απαλλαγή και διαρωτώ με μήπως συλλογικά στο μέλλον θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε αυτή η διαδικασία απαλλαγή να συμπεριληφθεί σε ένα έτο, να γίνει μάλλον μέσα σε ένα έτος. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ταβέρνα αν πιστεύει πω είναι δυνατόν να έχουμε του επαγγελμένου λογαριασμού όχι στα μέσα Ιουλίου όπω είναι σήμερα, αλλά να προηγηθεί αυτό τρει μήνες νωρίτερα. Αν γίνεται αυτό, όπω γίνεται εξάλλου και στι μεγάλου βιομηχανικού ελληνικού οποίο των οποίων ε, η χαρακτήρα των λογαριασμό δεν είναι περισσότερο πολύπλοκο από ότι οι δικοί μα λογαριασμοί. Τώρα, προλογαριασμοί 31 Δεκεμβρίου 2008, ε, δηλαδή στο φουλ της κρίσης. Αυτή η κρίση έχει επιπτώσεις στους λογαριασμούς. Και έπειτα, άκουσα τις παρατηρήσεις για τα ερωτήματα που τέθηκαν πέρσι. Για το αρνητικό αποθεματικό. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο Ταβέρν και τις υπηρεσίες του ποιες ήταν οι τεχνικές για να έχουμε καλύτερες ανταλλαγές για αυτό το θέμα. Εγώ σας λέω ειλικρινά ότι δεν μπορώ να αποφασίσω να έχω παγιωμένους λογαριασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό αποθεματικό γύρω στα 50 δις ευρώ. Δεν το έχω μαζί μου τον αριθμό. Τώρα, η εφαρμογή της αρχής ε, της ε, σύνεσης. Ε, καταγράφουμε το χρέος απέναντι στο προσωπικό, αλλά όχι την πίστοση προς τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν είμαι τεχνικός στο επίπεδο αυτό, αλλά πάντως δεν με πείθει. Δεν ξέρω γιατί. Και βρίσκω ότι η αρχή της σύνεσης για τα κράτη-μέλη... Εντάξει, τα κρατη είναι φερέγγι χρεώστες. Ωστόσο, ακούμε εδώ και εκεί διάφορες, ε, διάφορα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Εγώ θα ήθελα υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται μέσα εδώ, δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να πληρώνουν τη συντάξη του προσωπικού, θα πρέπει αυτό να συμπεριλαμβάνουν τους λογαριασμούς και μάλιστα μου φαίνεται πως είναι παράξενο ότι τα αποθυματικά για, τα, για το προσωπικό είναι 11%. Όχι μόνο δεν τα επιστρέφουμε, αλλά τα, δεν τα κρατούμε, αλλά τα επιστρέφουμε στα κράτη-μέλη. Τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτά που αντιστοιχούν στο προσωπικό. Εγώ λοιπόν υποβάλλω την ιδέα, κύριε Πρόεδρε, να γίνει, να σκεφτούμε την ύπαρξη ενό συνταξιδοτικού ταμείου, ώστε να υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη να καταβάλουν αυτά τα ποσά. Είναι 40 δι ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση 4 δι από χρόνο σε χρόνο και τα κράτη-μέλη δεν είμαι βέβαιο τι κάνουν. Εγώ πάντω θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανακτά αυτά τα ποσά. Για να μιλήσω τώρα για το Γαλιλαίο υπάρχουν δύο πτυχέ, δηλαδή η έρευνα να κρατά τους λογαριασμού. Φυσικά όταν πρόκειται για ερευνητικέ δαπάνε, ε, δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν αυτά ε, τα ποσά, αλλά το να περιμένουμε οποιοδήποτε απογραφή για να καταγράψουμε το Γαλιλαίο που μας ανήκει μετά από τι πολιτικέ διαπραγματεύσει, πιστεύω πω ε, η λογιστική του μετάφραση θα μπορούσε να γίνει εκ νέου. Τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εγγύησεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από όσο γνωρίζω, αυτές οι εγγύησεις δεν ανταμείβονται. Στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είχα ζητήσει να ανταμείβονται αυτές οι εγγυήσει και ε, πώς αυτές καταγράφονται στους λογαριασμούς και μήπως θα πρέπει αυτό να γίνεται με βάση μια έμεση επιδότηση που δίνουμε στην ε, ΕΤΕ σε περίπτωση ε, αποζημίωσης. Πρόκειται για 100 ή 200 δις ευρώ. Είναι σημαντικά ποσά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέας. Η κυρία Μαρόν Ανδρέας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταβέρν που έκανε αυτή την παρουσίαση για του λογαριασμού. Διερωτώ με γιατί υπογράφει του λογαριασμού από τη στιγμή που δεν ήταν υπεύθυνο για τι συναλλαγές για το 2009. Και ήταν ο κύριο Γκρέι που ήταν υπεύθυνο για τι ε, διάφορε συναλλαγέ. Πάντω, ε, όσον αφορά ε, του λογαριασμού, ενεργητικό και παθητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπω ότι η προχρηματοδότηση έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η προχρηματοδότηση είναι χρήματα τα οποία έχουν φύγει από το λογαριασμό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ταβέρνα να μας εξηγήσει γιατί αυξήθηκαν αυτά τα ποσά και επίσης αν είναι ικανοποιημένο από την ε, πληρότητα του των στοιχείων αυτών. Γιατί τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Σταβέρνη τη Κομισιόν για να απαντήσει στα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν για την ανάκριση. Αναφέρομαι στο σημείωμα 6 των λογαριασμών που δίνει λεπτομέρειες, ίσως και υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες, για τα ποσά των οποίων η ανάκτηση έχει αποφασιστεί μέσα στο 2008. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για την ανάκτηση των διαστατικών ταμείων δεν μπαίνουν πολλά πράγματα στους λογαριασμούς, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου αυτές οι διορθώσεις γίνονται από τα κρατημέλη και ε, χορηγούνται σε άλλε δαπάνε από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αυτά όλα αναφέρονται στα σημειώματα λοιπόν, αλλά δεν εμπίπτουν, δεν εντάσσονται μάλλον στους λογαριασμού τη Ένωση. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, ο αριθμός που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε, που είναι μάλλον οι αριθμοί που μα έδωσε η κυρία Γκρέσλε και που σχετίζονται με τι δύο μεγάλε περιόδου για τι οποίε έχουμε δαπάνε στον προπολογισμό, παρουσιάζουν ε, ποσά τα οποία έχουν ανακτηθεί αλλά που είναι αντικείμενο διορθώσεων ε, χρηματοπιστωτικών χωρίς απόφαση της Κομισιόν σε ένα μεγάλο τους ε, μέρος και αυτό εξηγεί ίσως την σύγχυση που μπορεί να προκληθεί από την ανάγνωση αυτών των σημειώσεων. Ναι, αν μεταφέρονται οι προπολογισμοί και αν, συγγνώμη, αν μεταφράζονται οι λογαριασμοί, ναι, μεταφράζονται και στη δική μας γλώσσα, κύριε Ντί. Παγιωμένοι λογαριασμοί. Αυτοί προετοιμάζονται μέσα Ιουλίου. Ε, με ρωτάτε αν μπορώ να το κάνω τρεις μήνες νωρίτερα. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση επί τη βάση των προσωρινών λογαριασμών που ε, καταρτίζονται τέλη Μαρτίου και που, προφανώ, ε, που πιθανότατα μάλλον θα επέτρεπε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πεδίο μέχρι ότου να γίνει η συζήτηση και για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα μας επέτρεπε αυτό να έχουμε πιο εις βάθος μελέτη πριν μπουν στα, πρακτικά, στην ατζέντα μάλλον αυτής εδώ της Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε θεσμικό όργανο οφείλει να προετοιμάσει τους προσωρινούς του λογαριασμούς, ότι έπειτα τους υποβάλλουμε στο ελεγκτικό συνέδριο ώστε να το μελετήσει πριν να τα υιοθετήσουμε οριστικά. Τώρα, αν η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιπτώσει στους λογαριασμούς, θα έλεγα ναι. Και είναι και η απάντησή μου στην κυρία Ανδρέα Σένα όσον αφορά το ύψος της προχρηματοδότησης. Και γιατί αυτό. Γιατί ε, στα διευθυντικά ταμεία οι κοινοτικέ παρεμβάσει συγχρηματοδοτούνται. Πράγμα που προποθέτει φυσικά ότι τα κράτη ή οι περιφέρειε ή οι ιδιώτε εταίροι συχνά ε, καταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης. Συχνά η κοινοτική χρηματοδότηση είναι μικρότερη από το 50%. Η κρίση και η ανάγκη των κρατών να κινητοποιήσουν ε, σημαντικά ποσά και συγκεκριμένα για να λύσουν την χρηματοπιστωτική τους κρίση, ίσως, και λέω ίσως, να αποτέλεσε έναν παράγοντα για το γεγονό ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των διαφόρων προγραμμάτων, άρα λιγότερε δαπάνε. Οι προχρηματοδοτήσει αυξάνονται διότι δεν καταναλώνονται. Και άρα τα χρήματα που καταβάλλονται παραμένουν προχρηματοδότηση. Και σίγουρα είναι αυτή η εξήγηση που οδηγεί στο ότι οι προχρηματοδοτήσει είναι πολύ υψηλέ στο τέλο του 2008. Μειώνονται όμω το 2009 και στου λογαριασμού του 2009 θα έπρεπε να έχουμε κανονικά λογαριασμού που θα είναι κάπω διαφορετικοί υπό αυτή την έννοια. Και σα θυμίζω ότι είμαστε ακόμα στι αρχέ του Νοεμβρίου. Το θέμα του αρνητικού αποθεματικού το έχουμε συζητήσει επί μακρόν, κύριε Οντή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από να εφαρμόσω τα διεθνή, τις διεθνείς προδιαγραφές για το δημόσιο τομέα, γιατί διαφορετικά θα με επέκρινε το ελληνικό συνέδριο, οι αρχές της αρμόδιας επί της απαλλαγής, πράγμα το οποίο κανείς δεν το επιθυμεί. Και άρα λοιπόν εγώ τηρώ τους κανόνες ε, Έχουμε μία λογιστική σύμβαση. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε πίστοση ε, σε έναν προπολογισμό μια πίστοση που δεν είναι πραγματική πίστοση. Μια εγγύηση γίνεται ε, ε, απτή και εγγράφεται από τη στιγμή που ε, χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για το Συνταξιδιωτικό Ταμείο και για το ΦΕΑΓΑ, αλλά είναι μια σύμβαση. Αυτό δεν αναιρεί τίποτα από την εγγύηση που δίνουν τα κράτη-μέλη. Το θέμα του Ταμείου Συνταξιοδότηση νομίζω πω σα είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Το έχουμε μελετήσει κατά τη διάρκεια τη τελευταία μεταρρύθμιση του ε, καταστατικού εργασίες στις οποίες συμμετείχα και θα πρέπει να σας πω ότι αυτό προσκρούει σε τεράστιες δυσκολίες. Θα πρέπει επίση να δούμε πώς θα επενδύσουμε αυτό το ταμείο, πώς θα το διαχειριστούμε και υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων δεν είμαι βέβαιος πώς θα έχουμε ε, κάθε εγγύηση ώστε αυτή είναι η καλύτερη λύση και η πιο ασφαλής από ότι μια ε, χρηματοδότηση αλληλέγγυα την οποία εγγυώνται τα 27 κράτη-μέλη. Τώρα για τον Γαλιλαίο η μεταφορά ε, της κυριότητας είναι αυτή που θα οδηγήσει στην εγγύηση. Ε, θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει για τους λογαριασμούς 2009, αλλά όχι για το Γαλιλαίο. Θα είναι το 2010 αυτό και ίσως και το 2011. Όσον αφορά τις εγγύησει για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ΕΤΕ, είναι στοιχεία εκτός προπολογισμού που βρίσκονται στη σελίδα 87 ε, των σημειώσεων για 17 δις. Είναι διαθέσιμα τα ποσά, είναι διαφανή και οι συμφωνίες ε, θέλουν αυτές οι πληροφορίες να βρίσκονται στις σημειώσεις και όχι στους λογαριασμούς. Η κυρία Αντρεσέν με ρωτά γιατί εγώ υπέγραψα τους λογαριασμούς ενώ ο κύριος Γκρέι ήταν αυτός ο οποίος έκανε τους προσωρινούς λογαριασμούς. Ναι, εκείνος υπέγραψε ο κύριος Γκρέι τους λογαριασμούς της 21η Μαρτίου και μετά εγώ τους δέχτηκα αφού επιμακρό συζήτησα μαζί του για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκαν αυτοί οι λογαριασμοί και είχα κάθε διαβεβαίωση πως αυτοί οι προσωρινοί λογαριασμοί καταρτίστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες και υπέγραψα τους οριστικούς λογαριασμούς μετά από κάποιες διορθώσεις ανάμεσα στην προσωρινή και στην οριστική βάση όπως αυτή αυτό ε, προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Απάντησα ήδη για το θέμα της αύξησης των προχρηματοδοτήσεων. Βασικός λόγος είναι ότι τα χρήματα αυτά προκαταβάλλονται στα κράτη-μέλη και δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες στις οποίες να μπορούμε να καταγράψουμε στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων. Και γι' αυτό και το οικονομικό μας αποτέλεσμα είναι, είναι πολύ ψηλό φέτος. Εγώ είμαι ε, ικανοποιημένο σε λογικό βαθμό για όλα τα σημαντικά στοιχεία όπως σας το ε, υπέγραψα και δεν έχω λόγο να αμφισβητώ την υπογραφή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά δύο ερωτήσεις θέλω να ξαναδιατυπώσω γιατί δεν απαντήθηκαν πιστεύω και δεν θέλω να κάνω τον ξέρω, αλλά παρόλα αυτά στην προχρηματοδότηση ξέρουμε από την έκθεση του συνεδρίου ότι στις πληρωμές διαθετικό Ταμείο για το 2008 από 11,8 δις 11,7 ήταν προχρηματοδοτημένα κονδύλια. Το πρόβλημα λοιπόν της προχρηματοδότησης είναι πολύ σοβαρό. Και όταν ξέρει κανείς και η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολισμού έδωσε μάχη κατά της αλλαγής των κανόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή προχρηματοδότηση κατά 100%. Αυτά δεν είναι προχρηματοδοτήσεις πλέον, αλλά είναι ε, εξαποκοπής ε, πληρωμή η καταποκοπή πληρωμή ευθύ εξ αρχή για ένα σχέδιο. Ε, τότε λοιπόν πιστεύω ότι τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε του χρόνου τίθενται, ε, στο μέλλον τίθενται επί τραπέζης. Αυτό ήθελα να αναφέρω για την προχρηματοδότηση ως πρόβλημα. Έχουμε υπόψη την προχρηματοδότηση, διότι θα έχουμε το αυριανό πρόβλημα μπροστά μας που πρέπει να αντιμετωπιστεί και σκεμμένα και ηθελημένα και σίγουρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξετάσουμε σε βάθος προσεκτικά όπως πρέπει. Τώρα για την ανάκτηση κονδυλίων θέλω να ξαναθέσω το θέμα. Θέλω και πάλι να ξαναρωτήσω. Σίγουρα σας διέφυγε, α και γι' αυτό θα πρέπει να απαντηθεί. Το νέο σχήμα για την ανάκτηση που με το ελεγκτικό συνέδριο θα προωθηθεί, κατά πόσο έχει οριμάσει. Μπορεί κάποιος από το ελεγκτικό συνέδριο να πει κατά πόσο αυτό το σχέδιο έχει προχωρήσει και κατά πόσον θα έχουμε αξιόπιστα ποσά για ανάκτηση. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Για να έχουμε κάποια τάξη όσον αφορά τα θέματα ανάκτηση. Και αυτό είναι θέμα κλειδί για μας. Δεν μπορούμε με 10 περίπου 12% αχρεωστήτως καταβληθέντα κονδύλια στα διαθετικά ταμεία να πούμε ότι ικανοποιούμαστε. Είναι 12 δις Είναι σημαντικό το ερώτημα. Τι ανακτάτε από αυτό το ποσό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα για μας. Για μας θα ήταν πρόοδος αν είχαμε στατιστικά στοιχεία που θα μας δίνατε ανακράτος μέλος ως κλίδα Πόσα δηλαδή τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ανακτήσουν και πόσα πραγματικά ανέκτησαν σε, ε, όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Θα ήταν πρόοδο για μα κάτι τέτοιο και γι' αυτό παράκλησή μου. Τέτοια στατιστικά στοιχεία θα μπορούσατε να μα τα διαθέσετε, να συντάξετε ένα τέτοιο κατάλογο και να μα τον διαθέσετε. Διότι θα μα βοηθούσε φυσικά το πρόβλημα τη ανάκτηση πολύ πιο στοχοθετημένα να το αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δεν πρέπει με ισοπεδωτικό τρόπο όλοι να αντιμετωπίζονται ισοπεδωτικά. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα για το πρόβλημα που υφίσταται στην ίδια την έδρα ενό κράτου μέλου. Πού υφίστανται τα προβλήματα προβλήματα. Θα θέλαμε ένα κατάλογο τι έχει γίνει και κατά πόσο έχουμε προχωρήσει. Και στατιστικά στοιχεία ανά κράτο μέλο, όπου θα αναφέρεται τι γίνεται για τα, με τα κράτη-μέλη για αυτό το φαινόμενο το οποίο σχεδιαγραφήθηκε. Δηλαδή, μετάθεση των κονδυλίων μέσα σε σχέδια, σε άλλα προγράμματα και έτσι πρέπει να δούμε και να ανοιχνεύσουμε τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ντί παρακαλώ. Πολύ σύντομα, όσον αφορά τι ε, εγγύσει, είδα τα 17 δισεκατομμύρια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εδώ πέρα αναφερόμαστε όμω στην πληρωμή των εγγύσεων. Για τι ε, χρηματοοικονομικέ αγορέ μιλάμε για ένα ποσοστό 0,5-1%. Επομένω, ε, για τα δικά μα ποσά μιλάμε για περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει λοιπόν μία απώλεια πόρων δεν υπάρχει πάντω κάπω ένα πρόβλημα. Απλώ αυτό που θα ήθελα να γνωρίσουν είναι αν αυτή την απώλεια την καταγράφουμε στον προπολογισμό ή όχι. Ή αν πρόκειται για μία έμεση χρηματοδότηση, επιδότηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε προχρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση, για την προχρηματοδότηση. Αυτή δεν επηρεάζει τον, το βαθμό της παρέμβασης που γίνεται στις δαπάνες. Η συγχρηματοδότηση καταγράφεται όμως στις βασικές πράξεις και τι σημαίνει ότι η κοινοτική παρέμβαση ε, έχει ένα πλαφόν. Χρησιμοποιούμε δηλαδή κάποια ποσά τα οποία έχουν προχρηματοδοτηθεί. Από τη μια λοιπόν έχετε μία εκταμείευση ενώ από την άλλη έχετε απλω μία καλύτερη παρουσίαση των δαπανών. Όσον αφορά την ανάκτηση, αναφερθήκατε στο ποσοστό του 10-12%. Είναι το ποσοστό σφάλματος το οποίο έχουμε στην έκθεση του 2007 για τα διαφορετικά ταμεία. Τι σημαίνει αυτό. Το λεκτικό συνέδριο εδώ πέρα είδε ότι υπάρχει αυτό το σφάλμα αυτό το ποσοστό σε ένα δείγμα δαπανών των διεθνωτικών ταμείων για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι για ένα κράτος μέλος, ούτε για ένα σύνολο κρατών μελών, ούτε ξερώντας το ένα ή το άλλο μέρος κράτος μέλος. Είναι μία δειγματολογική ανάλυση που γίνεται αντιπροσωπευτική σε επίπεδο όλων των κρατών μελών και όχι για ένα κράτος μέλος ή για μια συγκεκριμένη ομάδα κρατών μελών. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στην ετήσια έκθεση των διαρθρωτικών ταμείων. Εκεί πέρα μπορείτε να δείτε ποσοστά σφάλματο και δαπάνε για κάθε κράτο μέλο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε όμω από το ελεκτικό συνέδριο να κάνει κάτι τέτοιο. Το ελεκτικό συνέδριο αυτό το οποίο κάνει είναι ότι λαμβάνει κάποια δειγματοληπτικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη και κάνει μια έκθεση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ για τα όσα είπατε με το ζήτημα της ανάκτησης, προσπαθούμε να βελτιώσουμε το ζήτημα αυτό. Είπατε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη περισσότερο τις δράσεις εσωτερικού ελέγχου και στις 28 Οκτωβρίου υπέβαλε μια σχετική έκθεση και μια ακόμα προβλέπεται για τις αρχές Ιανουαρίου όσον αφορά την δηλαδή, τον εσωτερικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχετε λοιπόν την δυνατότητα να δείτε και στα πλαίσια του ελέγχου αυτού πώς συμπεριφέρεται το κάθε κράτος μέλος στα πλαίσια των διευθυντικών ταμείων. Εμείς όμως σε επίπεδο ενοποιημένων λογαριασμών μιλάμε μόνο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Κύριο Ντί, φοβάμαι ότι ε, όντως κάνουμε ένα δώρο αυτή τη στιγμή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την πληρωμή των εγγύησεων. Πρόκειται για μία σύμβαση, πρόκειται για μία συμφωνία νομική που είχε ληφθεί στο παρελθόν και δεν μπορούμε εμείς να δράσουμε από αυτού ή να επιφέρουμε μια αλλαγή ως εκτελεστική επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ανδρεάσεν. Σας ευχαριστώ. Εγώ επανέρχομαι στη Χρηματοδότηση και επιστρέφω την προσοχή σα στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύει το 45% του ενεργητικού και 33% του προπολογισμού. Δεν μπορώ να δεχτώ τη, τα όσα μας λέει ο κύριο Ταβέρνα, ότι δηλαδή η προχρηματοδότηση δεν έχει σχέση και δεν έχει επιπτώσει στι δαπάνε. Ε, είναι δαπάνες οι οποίες έχουν ε, καταβληθεί εκ των προτέρων και πρέπει να προσέξουμε ώστε να έχουμε την τεκμηρίωση που να επαληθεύει πως τα χρήματα αυτά έχουν ε, δαπανηθεί σωστά. Είναι τεράστια ποσά τα οποία δαπανώνται σε τομείς όπου το, δικαστη... το ελεγκτικό συνέδριο έχει βρει τον υψηλότερο βαθμό σφαλμάτων, δηλαδή διορθωτικά ταμεία και ε, αγροτική ανάπτυξη, μάλλον ανάπτυξη υπαίθρου. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έτσι ελαφρύ την καρδία να πούμε πως δεν ε, επηρεάζει αυτό τις δαπάνες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, μία ή άλλη σκέψη που υπήρξε. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Όμως, θέλω να επισημάνω, εκείνος ο οποίος προσπαθεί τον έλεγχο προϋπολογισμού να τον κάνει σοβαρά, <clears throat> είναι δυστυχισμένος ταλέπορος κάνω λόγο για μένα, την ίδια για παράδειγμα, γιατί το, τι βρίσκει κανείς ε, ως ποσό, σε ποιο έγγραφο και που κάτι τυχαία ε, δημοσιεύθηκε, δημοσιοποιήθηκε ή όχι, για παράδειγμα για το Διαθετικό Ταμείο 2008, αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο μας υπέρμετρα. Τώρα για την έκθεση της ετήσιας ε, ε, έκθεσης δραστηριοτήτων σε σχέση με τα αγροτικά υπάρχει πράγματι στατιστικός καταλόγος για τα ποσοστά σφάλματος ανακράτος μέλος. Αν μπορώ να βρω αυτό τότε μου αξίζουν συγχαρητήρια γιατί είναι κρυμμένο σε κάποια σελίδα. Τώρα Πού να βρω τα άλλα στοιχεία τα οποία ζητώ. Για παράδειγμα, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων έχει εύρος 3.000 σελίδων και παραπάνω. Κάποιος, κάθε εισηγητή για την χορήγηση απαλλαγή ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Βρίσκονται πληροφορίε θαμμένε μέσα σε αυτέ τι χιλιάδες σελίδε. Και σε σχέση με την πιο αποτελεσματική μέθοδο να σκοτώνει κανεί ευρωβουλευτέ με όγκο χαρτιού, με όγκο εντύπων, είναι μία μέθοδο θα έλεγα, αποτελεσματική. Αυτό που θέλω είναι μια επισκόπηση για την ανάκτηση. Γι' αυτό θερμή παράκληση. Ω μικρή Ευρωβουλευτήνα εναντί, εναν, εναντί ενό μεγάλου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, να μα βοηθήσετε παρακαλώ, να μα δώσετε αυτέ τι πληροφορίε από ταμείο σε ταμείο, ανά ταμείο, ώστε να ξέρουμε από κράτο μέλο σε κράτο μέλο τι γίνεται, να ξέρουμε πού υπάρχουν τα προβλήματα. Θέλω να παρακαλέσω τον συνάδελφο Λιμπεράτσι αυτή αυτό το αίτημα να το συμπεριλάβει στην έκθεσή του λέξη προ λέξη κυριολεκτικά. <clears throat> Αν δεν μπορέσουμε να θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα για να έχουμε μια καλώ λειτουργούσα διοίκηση και πρέπει να βοηθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να διαδραματίσουν το ρόλο του, να μεριμνήσουν για τη σωστή εκτέλεση δηλαδή και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Δείξτε κατανόηση για μένα παρακαλώ. Με την απάντηση κάπω αμήχανη είμαι και δεν είμαι ικανοποιημένη ιδιαίτερα. Υπάρχουν τόσα πολλά έγγραφα, γι' αυτό θερμή παράκλησή μου. Αυτά τα στοιχεία να μας τα δώσετε για κάθε ταμείο ξεχωριστά, για κάθε κράτος μέρος ξεχωριστά. Σε ένα ξεχωριστό φυλάδιο, σε ξεχωριστές σελίδες που θα τυπωθούν αυτά άσχετα που και πώς, αλλά θα πρέπει όλες οι πληροφορίες σε ένα σημείο να είναι προσπελάσιμες, προσβάσιμες για μα. Αυτό νομίζω ότι θα ε, αντιμετωπιζόταν και και ικανοποιητικά από το ελεγκτικό συνέδριο που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ σύμφωνα με τις προσδοκίες ε, πρέπει να πω ότι έχουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά τα διαθωτικά ταμεία και όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Θέλω να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και να πω το εξής. Είναι έτοιμά μας αυτό. Ιδιαίτερα πρόκειται για την απλούστευση, την πιο απλή διάταξη και ρύθμιση των προγραμμάτων σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Έχουμε διάφορα προγράμματα και όσον αφορά την ευθύνη των κρατών μελών που επομίζονται την εκτέλεση αυτών. Πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν, μια και εξ ονόματός τους έχουν, ε, πρέπει να δημιουργήσουν μια σαφήνεια στο χρηματοδοτικό πλαίσιο από πλευράς τους και να έχουμε τα έσοδα τα οποία θα αναφέρονται σαφώς και την προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Να γίνει κάτι επιτέλους. Ε, εκεί να επικεντρωθούμε με ιδιαίτερο τρόπο. Και για τον περιορισμό των κονδυλίων ή των προϋπολογισμών δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι τελευταίοι αποδέκτες ε, αυτά τα κονδύλια τα έχουν πράγματι λάβει. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσει κανείς ότι με τον χρόνο θα αυξάνεται αυτό το ποσοστό και αυτό το τμήμα. Θέλω να επανέλθω στο ερώτημα το οποίο διατυπώθηκε προηγούμενα. Αξιότιμε κύριε Γενικέ Διευθυντέ, Διευθυντά, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριε Κάλλας, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε στην πρόταση της κυρίας Γκρέσλε και γοργά να ανταποκριθείτε και να αναλυθεί αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει απειλή πράγματι να υπάρξει συσσόρευση αθρηστικά των μη ανακτώμενων, μη ανακτηθέντων ποσών όσον αφορά τα διαθωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Είναι το τελευταίο έτος θα έλεγα τώρα όπου μπορούμε σε αυτό να προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε και μπορούμε να αντιδράσουμε. Δώστε μου μια απάντηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ταβέρν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ύψο των προχρηματοδοτήσεων εξηγείται ευκόλω. Βρισκόμαστε στην αρχή μια νέα νομοθετική νομοθετικής περίοδου 2007-2013. Εδώ έχουμε την χρήση 2008, δηλαδή το δεύτερο έτος μιας πολύ μακρά περίοδου. Είναι απόλυτα φυσιολογικό λοιπόν σε αυτή τη φάση, στο πέρας αυτή τη χρήση, ο προπολογισμό να δείξει ότι έχουμε προχωρήσει πολύ σε προχρηματοδότηση των διευθυντικών πολιτικών που εκτείνονται στο διάστημα 2007-2013 ο χρόνος εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων είναι πολύ μακρύς. Αυτό είναι γεγονό. Στη συνέχεια, καταβάλουμε πολλές φορές 10 χρόνια μετά από την έναρξη μιας περίοδου τα υπόλοιπα των ε, προκαταβολών που έχουν δοθεί. Δεν έχουμε κλείσει εξάλλου ούτε το 2006 όσον αφορά τις πληρωμές. Σήμερα ακόμη το, το ελεγκτικό συνέδριο που θα εκφραστεί εντός ολίγου έχει πάρει ένα δείγμα από τα διευθυντικά ταμεία που, συν, που αποτελείται από, την, ε, από πληρωμές 2000 με 2006. Υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό κενό, ένα μεγάλο κενό όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία ανάμεσα στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, τη δεσμεύση και την εκτέλεση επιτόπου και μετά τον έλεγχο τη εκτέλεση που γίνεται βεβαίω μόνο μετά από την εκτέλεση. Είμαστε λοιπόν στα τέλη του 2008, αλλά είμαστε σε κάποιο ένα πρώιμο στάδιο τη εφαρμογή των αποφάσεων για τα διευθυντικά ταμεία για το 2007-2013. Σημειώνω ότι ε, υπερβολικά πολλές πληροφορίες είναι σαν να μην υπάρχουν και δεσμεύομαι να σας δώσω τα στοιχεία ανά ταμείο. Θα τα ψάξουμε εμείς για τις λογαριασμούς σας και θα σας τα διαβεβάσω τα στοιχεία αυτά. Κύριε Λιμπεράτσχη, οι κυβερνήσεις δεν συγχρηματοδοτούν έχουν δυσκολίες να βρουν συγχρηματοδότηση ίσως. Α, αυτό αποτελεί απειλή για τις προκαταβολές. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι προχρηματοδοτήσεις δεν θα ανακτηθούν. Τίποτα δεν μας επιτρέπει να πούμε κάτι τέτοιο σήμερα. Τίποτα δεν μας επιτρέπει να το πούμε τη στιγμή που αποφασίζονται ή που, που κλείνουν οι λογαριασμοί της, την 31η Δεκεμβρίου 2008. Πρόκειται για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και φυσικά για η εκτέλεση των προγραμμάτων εποπτεύεται με πολύ αυστηρό τρόπο και ξέρετε σε ποιο βαθμό το ελεγκτικό συνέδριο αποδίδει πρωταρχική σημασία σε αυστηρό έλεγχο, στον αυστηρό έλεγχο που βάζει Κομισιόν και αυτό σύμφωνα με τις βασικές πράξεις, δηλαδή τις αποφάσεις του Συμβουλίου που προβλέπουν ότι τα κράτη έχουν τη δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουν τα χρήματα τα οποία τα ίδια ανακτούν από προγράμματα που δεν είναι ικανοποιητικά. Δηλαδή ο έλεγχος δεν είναι μόνο από πλευρά τη Κομισιόν. Τα χρήματα τα οποία ανακτώνται δεν ανακτούνται από την Κομισιόν. Υπάρχει ένα σύνολο μέτρων μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης από πλευρά των κρατών μελών που προβλέπεται από τι βασικέ πράξει και στι οποίε η Κομισιόν δεν μπορεί βέβαια να τις παραβλέψει.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 Μόλις ήρθε και ο, και του Ελληνικού Συνεδρίου, ο κύριος Καλτέρα, ζήτησε ο κύριος Μπούζεκ να καθυστερήσουμε λίγο την ακρόαση. Έχουμε το χρόνο να τον ακούσουμε με ηρεμία, όπω θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Επίτροπο κύριο Κάλαση και τον εισηγητή κύριο, Λιμπεράσκη και θα ξεκινήσουμε μετά τη συζήτηση. Πριν να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο, τον κύριο Καλτέρα, εγώ την Παρασκευή, όπως είχαμε συμφωνήσει, έλαβα το ενεργασία του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Οικονομική Χρήση 2008 και θέλω να υπογραμμίσω προσωπικά ε, τους επένους μου για την εξαίρετη εργασία του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πολύ σημαντικές πληροφορίε που μα επιτρέπουν να δουλέψουμε αποτελεσματικά φέτος, να σκεφτούμε την ανάλυση την οποία έχει κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, για τις πιο κρίσιμες πτυχές ε, που μπορούμε να δούμε εδώ. Μια ανάλυση πολύ προσεκτική που αφορά τα διάφορα κεφάλαια δαπανών, διευθυντικά ταμεία, έρευνα, μεταφορές, ενέργεια, ε, τα, ταμεία που, τα κονδύλια που πάνε στα κρατημέλη, τα κονδύλια που πάνε σε άλλα κρατημέλη, σε άλλα κράτη μάλλον, ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια για τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και για το μέλλον οι εργασίες του ε, ελεγκτικού συνεδρίου θα είναι θεμελιώδους σημασίας όπως πιστεύω επίσης και η σημασία που δίνουμε στο να ε, ενεργεί το ελεγκτικό συνέδριο πλήρως ανεξάρτητο και αυτόνομο από την, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. θα πρέπει να δούμε, να, να ελέγχονται όλα τα κονδύλια που δαπανώνται. Ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεματζίστρης για αυτές τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις σας και τα ευγενικά σας λόγια. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά τιμή για μένα να έχω αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την εφαρμογή, την εκτέλεση του προπολογισμού για το οικονομικό το 2008 και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι η πρώτη ευκαιρία που έχω επίσημα να προσφωνήσω και να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας μετά τις εκλογές και να γνωρίσω τα μέλη, τα νέα μέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να δραχθώ αυτή τη ευκαιρία να συγχαρώ να συγχαρώ όλους σας για την εκλογή σας και εσάς ε, ιδιαίτερα κύριε Ντεματζίστρης για τον διορισμό σας ως ε, Πρόεδρο της Επιτροπής. Είναι μια ετήσια έκθεση και που έχει παραθεί και που είναι πολύ διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Το 2008 θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μνήμη εξαιτία των γεγονότων τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική χρηματοοικονομική κρίση που εξακολουθεί να έχει σημαντικέ επιπτώσει στα κράτη-μέλη και στον προπολογισμό τη Ένωση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι εκθέσει και οι γνώμε του, του συνεδρίου έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Τουλάχιστον για να υπενθυμίζεται το διαρκέ πρόβλημα στον τομέα τη δημοσιονομική διαχείριση, τα διαρκή προβλήματα και οι προσπάθειε που γίνονται για να αντιμετωπιστούν και οι προκλήσεις που απομένουν να αντιμετωπιστούν. Θα ξαναγυρίσω σε αυτά τα θέματα υστερότερα κατά τη διάρκεια της παρεμβασή μου μετά την παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της, ε, αυτής της ε, ετήσιας έκθεσης για εφέτος. Πράγματι έχουμε τέσσερα κύρια μηνύματα <clears throat> μέσα σε αυτή την έκθεση που δίνουμε. Πρώτο μήνυμα. Ε, οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αξιόπιστοι για δεύτερο συνεχές έτος. Δεύτερο μήνυμα. Το επίπεδο των ε, παρατυπιών ε, έχει μειωθεί συνολικά σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των βελτιώσεων που σημειώθηκαν στη διαχείριση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσης, αλλά το ύψος των παρατύπων αυτών πληρωμών παραμένει σχετικά υψηλό Δεύτερον, οι συστάσει ε, του ελληνικού συνεδρίου από τα προηγούμενα έτη σε σχέση με τα όσα πρέπει να γίνουν εξακολουθούν να ισχύουν. Και τέλος, η απλούστευση εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα που πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή, να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Επιτρέψτε μου σε κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα να μείνω λίγο περισσότερο. Πρώτον, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών. Για δεύτερο συνεχές συναπτό έτο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει γνώμη χωρί επιφύλαξη, ανεπιφύλακτα δέχεται του λογαριασμού και το συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί παρέχουν πιστή εικόνα για κάθε ουσιώδη πλευρά τη οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 και όσον αφορά και τι πράξει, ε, τι ταμιακτικέ ροέ κτλ που λήγουν κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι λογαριασμοί είναι τέλειοι, ή ιδανικοί και τα συστήματα που του παράγουν είναι αλάνθαστα. Στην πραγματικότητα το συνέδριο υπογραμμίζει ότι υπάρχουν αδυναμίε στα λογιστικά συστήματα ορισμένων γενικών διευθύνσεων τη Επιτροπή που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των δημοσιονομικών πληροφοριακών στοιχείων. Παρότι δεν υπήρξαν σημαντικά σφάλματα, ουσιώδη σφάλματα όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στου λογαριασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξετάζει με τη δέουσα προσοχή τα ζητήματα που σημαίνει το συνέδριο. Όσον αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα των λογαριασμών και των πράξεων είναι το δεύτερο κύριο μήνυμά μα, ότι το επίπεδο παρατυπιών έχει μειωθεί συνολικά κατά τα τελευταία έτη χάρη στις βελτιώσεις στην διαχείριση του προπολογισμού. Αλλά όμως εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά τα επίπεδα κινδύνων σε ορισμένου τομεί. Όπως και στα προηγούμενα έτη, έτσι και για το 2008, το Ελεκτικό Συνέδριο δίνει χωρίς επιφύλαξη την ε, έγκριστη γνώμη του για τα έσοδα και τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Εν τούτης, η εικόνα είναι ανάμεικτη. Παραμένει ανομοιογενής, μόλον ότι σημειώθηκαν ορισμένε μεταβολές από έτος σε έτος. Το συνέδριο διατυπώνει ανεπιφύλακτα, χωρί επιφύλαξη, άποψη για τι δαπάνε όσον αφορά την εκπαίδευση και την ιδιότητα του πολίτη και τι διοικητικέ και λοιπέ δαπάνε. Σε αυτού του τομεί το συνέδριο εκτιμά ότι το ετήσιο σφάλμα βρίσκεται κάτω από 2%. Για την παιδεία και την εκπαίδευση και για την ε, ε ηθαγένεια, την ιδιότητα του πολίτη, το γεγονό αυτό οφείλεται στο ότι εν πολύ στο μεγάλο αριθμό προπληρωμών το 2008 για τι οποίε ελάχιστε προποθέσει υπάρχουν και κατά συνέπεια επηρεάζουν πολύ λιγότερο από σε σύγκριση με ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές. Όμως τα, ε, τα συστήματα στον τομέα αυτό συνεχίζουν να αξιολογούνται μόνον όσο μερικώς αποτελεσματικά. Εξάλλου διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα στον τομέα των διοικητικών δαπανών ε, εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσει του δημοσιονομικού κανονισμού όπως και κατά προηγούμενα έτη. Για τη γεωργία και τους φυσικούς συνέδριο για πρώτη φορά διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ε, εξαιρουμένης της αγροτικής ανάπτυξης οι πολιτικές, οι πληρωμές ήταν από κάθε ουσιώδη πλευρά νόμιμες και κανονικές. Για πρώτη φορά το συνέδριο εκτιμά ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος για την εν λόγω ομάδα βρίσκεται κάτω από 2%. Μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Όμως εν τούτης, το εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος για το τμήμα των δαπανών που αφορά την γεωργική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της υπαίθρου, εξακολουθεί να υπερβαίνει το 2%, μολονότι είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Οι ανεπάρκειε στα συστήματα υποπτίας και ελέγχου που αφορούν την ανάπτυξη τη υπαίθρου συνέβαλαν σημαντικά στο να αξιολογήσει συνολικά το συνέδριο θετικά μόνο μερικώ αποτελεσματικά τα συστήματα που αφορούν τη γεωργία και του φυσικού πόρου. Μολονότι το συνέδριο διαπίστωσε ότι το ΟΣΔΕ είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την μείωση του κινδύνου παράτυπων δαπανών. Το συνέδριο διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη επίση όσον αφορά την ομάδα πολιτική οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων λόγω των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν στι πράξει που αφορούν <clears throat> το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Όσον αφορά τι ομάδε πολιτική συνοχή έρευνα, ενέργεια και μεταφορών και την εξωτερική βοήθεια ανάπτυξη και διεύρυνση, το συνέδριο θεωρεί, εκτιμά και εξακολουθεί να διατυπώνει αρνητικέ γνώμε, καταλήγοντα στο συμπέρασμα ότι επηρεάστηκαν από σιώδη σφάλματα σε διαφορετικά επίπεδα. Συνοχή. Η δεύτερη σημαντικότερη ομάδα, το περίπου 1 τρίτο του προπολογισμού. Είναι ο τομέα ο οποίο πλήττεται σημαντικότερα από σφάλματα. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι εκτιμά ότι 11% τουλάχιστον του ε, συνολικού ποσού που αποδόθηκε δεν θα έπρεπε να είχε εκταμιευτεί αχρεωστήτως λοιπόν. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όσον αφορά τα προηγούμενα έτη, τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν από το συνέδριο αφορούν ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές στα έργα ε, του τομέα συνοχής όσον αφορά την περίοδο 2000-2006. Σημαντικό τμήμα του εκτιμόμενου ποσοστού σφαλμάτων αφορά σφάλματα επιλεξιμότητας, παράδειγμα, χάρη σε ορισμένα έργα που δεν πληρούσαν τις ε, συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Η Επιτροπή απάντησε κατ' παρελθόν ισχυριζόμενη ότι οι μηχανισμοί διόρθωσης και ανάκτησης χρησιμεύουν για τη, στη μείωση των επιπτώσεων των σφαλμάτων που ανοιχνεύονται από το συνέδριο κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής. Όμως ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδείξει αφενός το εύρος αυτό διότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές δεν δίνουν πλήρη στοιχεία και αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τις διορθώσεις αυτές. Και επειδή είναι <clears throat> πρώιμο το στάδιο μέτρησης επιπτώσεων εν εξελίξει δράσεων για να δει κανείς το τι γίνεται σε σχέση με τη διαχείριση διαθωτικών ενεργειών. Επιπλέον, το ελεγκτικό συνέδριο επεσήμανε περιπτώσεις αντικατάστασης από τα κράτη-μέλη των μη επιλέξιμων δαπανών με νέες δαπάνες, οι οποίες ε, ήταν επίσης μη επιλέξιμες <laughs> λόγω ανεπαρκούς εκπροτέρων, ελέγχου, εξάντε ελέγχου. Στην έκθεση παρατίθεται, το παράδειγμα μιας διαχειριστικής αρχής που αντικατέστησε ένα έργο του ΕΤΠΑ και που είχε απορρίψει απορρίψει η Επιτροπή με ένα άλλο έργο για το οποίο οι δηλωθήσει δαπάνε ανήλθαν σε 5,7 εκατομμύρια και το οποίο ήταν επίση μη επιλέξιμο διότι είναι γνωστό ότι το σχέδιο αυτό είχε καθοριστεί με τρόπο που δεν μπορούσε να εγκριθεί. Το έργο όσον αφορά την περίοδο τώρα 2007-2013 όλε οι πληρωμέ, οι περισσότερε πληρωμέ είναι προχρηματοδοτούμενε και υπάρχουν ε, σχετικά περιορισμένε προποθέσει για αυτέ. Είναι συνεπώ πολύ πρόημο το στάδιο αυτό να κρίνουμε αν οι αλλαγέ στου κανόνε. ή στα συστήματα εποπτείας και επιτήρησης για το 2007-2013 ως περίοδο είχαν θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των επιπέδων σφαλμάτων στις ε, ε, προπληρωμές και στις ενδιάμεσες πληρωμές. Ωστόσο το συνέδριο ενοχλήθηκε και με ανησυχία σημείωσε τις καθυστερήσεις όσον αφορά τις εγκρίσεις ε, από τα κράτη-μέλη, μια και έχουν επιβραδύνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων όσον αφορά την ανείχνευση το, αυτών στο στάδιο έναρξη Κατά τέλη του 2008 σε 38% των περιπτώσεων τα κράτη-μέλη υπέβαλαν αυτά τα ε, έγγραφα με καθυστέρηση στην Επιτροπή. Όσον αφορά την ε, έρευνα, την ε, ενέργεια και τις μεταφορές, μολονότι η ομάδα πολιτική εξακολουθεί να επηρεάζεται από σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων, το συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησαν στη μείωση των σφαλμάτων. Όπω και κατά το παρελθόν, τα σφάλματα που ανοιχνεύτηκαν αφορούν κυρίω στην την απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών και προσωπικών και μέσων δαπανών για τα ερευνητικά έργα. Μία από τι αιτίε των σφαλμάτων αυτών απαιτεί το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο και το μεγάλο αριθμό περίπλοκων κριτηρίων επιλεξιμότητα συμπεριλαμβανομένη και τη απέτηση για παροχή αποδείξεων. Το συνέδριο έκρινε λοιπόν ότι τα συστήματα ελέγχου είναι εν μέρη μόνο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, <clears throat> οι δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται από πλευρά δικαιούχων πρέπει να, ελέγχονται, να συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό ελέγχο εκδιδόμενο από ανεξάρτητο ελεγκτή. Εν τούτης όμως, στο ίμιση και παραπάνω σχεδόν από τις περιπτώσεις αυτές όπου το συνέδριο διαπιστώνει σφάλματα στις δηλώσεις δαπανών, αυτές είχαν πιστοποιηθεί χωρίς επιφύλαξη. Επιπλέον, παρά την σημαντική αύξηση της κάλυψης ε, των καταστατικών ελέγχων από την Επιτροπή, το ύψος των ανακτήσεων που είχαν δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2008 ήταν χαμηλό και δεν είχαν επιφύλαξη επιβληθεί κυρώσει. Για την ομάδα πολιτική εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη και διεύρυνση, το συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πληρωμέ επηρεάστηκαν από σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων. Όπω και κατά τα προηγούμενα έτη, το συνέδριο εντόπισε περιπτώσει μη επιλέξιμων δαπανών, έλλειψη δικαιολογητικών και παρατυπιών στι διαδικασίε σύναψη συμβάσεων. Διαπιστώθηκε εκ νέου ότι τα συστήματα που εφαρμόστηκαν από τι αρμόδιε γενικέ διευθύνσει ήταν μόνο μερικώ αποτελεσματικά, αλλά για διαφορετικού λόγου εκάστοτε. Εξακολουθούν να εντοπίζονται σε επίπεδο φορέων υλοποίηση και αντιπροσωπιών παρά σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών για την εξωτερική βοήθεια και για την αναπτυξιακή βοήθεια οι οποίε χρηματοδοτούνται επίση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Σε άλλου τομεί οι ανεπάρκειε που σημειώθηκαν αφορούσαν κυρίω πτυχέ των καταστατικών ε, δράσεων και του εσωτερικού ελέγχου. Συνολικά τα ποσοστά σφαλμάτων φαίνεται ότι μειώνονται χάρη στι βελτιώσει που έχουν επιτευχθεί στην διαχείριση του αλλά τα νομικά πλαίσια εξακολουθούν να είναι πολύπλοκα και περίπλοκα και τα προβλήματα παραμένουν σε ορισμένα συστήματα ελέγχου. Τώρα, τίθεται το εξή ε, ε, ζήτημα. Ε, το ερώτημα με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί περαιτέρω το επίπεδο των παράτυπων πληρωμών. Και η απάντηση που δίνει το ελεγκτικό συνέδριο περιλαμβάνει δύο παραμέτρους. Περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου όσον αφορά τη διαχείριση και κατά περίπτωση εκάστοτε απλούστευση των κανόνων και των κανονισμών. Αυτό με οδηγεί τώρα στο τρίτο κύριο βασικό μήνυμα τη έκθεσή μα. Βελτίωση δηλαδή τη αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτεία και ελέγχου. Οι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου από τα προηγούμενα έτη σε σχέση με το πώ μπορούν να βελτιωθούν τα συστήματα συστημικά εξακολουθούν να ισχύουν πρέπει να ε, θεωρούνται ως μέρος μιας ε, ενρευστό ενεξελίξη διαδικασία, στο πλαίσιο τη οποία θα απαιτηθεί χρόνο έω ότου καταστεί δυνατό να θεωρηθούν αποτελεσματικά τα σχετικά αυτά μέτρα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα κατά προτεραιότητα οι συγκεκριμένε αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από συνέδριο, πολλέ από τι οποίε, μόλι σας χειαγράφησα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ξεχωριστά στη συνέχιση τη βελτίωση των μηχανισμών διορθωση των σφαλμάτων μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων και προβλέποντας ε, το κλείσιμο των, της περίοδου 2000-2006 επιπλέον και παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την βελτίωση της εποπτείας πρόσφατα Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί επιπρόσθετα να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά λοιπόν ε, το Ελληνικό Συνέδριο στην Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλιστεί και να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτείας και ελέγχων. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της ε, συνεκτικότητας και των αξιολογήσεων όσον αφορά τα ε, συστήματα εποπτείας και ελέγχου που περιλαμβάνονται στι αιτήσει εκθέσει δραστηριοτήτων και τι δηλώσει βελτίωση τη διατύπωσης σε αυτές των επιφυλάξεων καθώ και τη βελτίωση ε, τη ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών σε σχέση με τι δημοσιονομικέ διορθώσει και ανακτήσει. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να επιζητεί την αποκόμιση βεβαιότητα, ε, δήλωση αξιοπιστία από τι ε, ετήσιες συνόψει και τις εκ των προτέρων δηλώσει όλων των κρατών μελών καθώ και από τι εθελοντικέ πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουν, αναλαμβάνουν ορισμένα κράτη-μέλη με τη μορφή εθνικών δηλώσεων ή ανώτατα όργανα ελέγχου πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο πλαίσιο αναφορά όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματο, ε, τι ε, δημοσιονομικέ διορθώσει και τι ανακτήσει, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι δράσει που θα αναλαμβάνονται θα είναι πιο αποτελεσματικέ για την εποπτεία και ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τη μελέτη σχετικά με το κόστο και όφελο, την αναλογία κόστο-οφέλου στου διάφορου τομεί ε, πολιτική. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση, ο εντοπισμό των τομέων όπου θα μπορούσαν να επιτευχθούν περισσότερο με τι υπάρχουσε δαπάνε, τι διαθέσιμε δαπάνε και του ελέγχου και ο εντοπισμό περιπτώσεων στι οποίε. Ε, είναι αδύνατη η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ του κόστους και, του ε, και ελέγχων και του ωφέλους ε, που επιτυγχάνεται. Στο πλαίσιο των εν λόγω αυτών αναθεωρήσεων, οι νομοθετικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσουν πώς μπορούν να επαναπροσδιοριστούν τα συστήματα ελέγχου με γνώμονα τις υλοποιήσεις και όχι τόσο τις εισρωές. Με άλλα λόγια, αντί να προσδιορίζεται ο αριθμός ελέγχων προς διενέργεια, στόχος πρέπει να είναι ο καθορισμός ε, ενός επίπεδου εναπομένοντος κινδύνου παρατυπιών που δεν πρέπει να υπερβαίνει το συστημικό ε, ποσοστό κινδύνου όσον αφορά το ανεκτό ε, επίπεδο σφάλματος. Ωστόσο υπάρχουν όρια στη μείωση του επίπεδου των παρατυπιών που μπορεί να επιτευχθεί ε, το επίπεδου των παρατυπιών που μπορεί να επιτευχθεί ως επίπεδο μέσω της βελτίωσης αποτελεσματικότητας των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου. Ας αναφέρουμε εδώ την ε, διαρκή ανάγκη για απλούστευση. Σε πολλούς από τους τομείς όπου το ελεγκτικό συνέδριο συνεχίζει να διαπιστώνει υπερβολικά υψηλό επίπεδο σφαλμάτων, αιτία των σφαλμάτων είναι τα υπερβολικά πολύπλοκα αυτά πλαίσια και οι κανόνε, οι περίπλοκοι κανόνε και οι κανονισμοί. Συνεπώ, η απλούστευση εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Όπω υπογραμμίζουμε από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου στη δήλωση αξιοπιστία, οι τομέί όπου εντοπίζονται υπερβολικά υψηλά επίπεδα σφαλμάτων είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκού ή ασαφεί ε, νομικού κανόνε και απαιτήσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην απλούστευση στου ε, τομεί αυτού. Όπω συχνά έχει τονίσει το ελεγκτικό συνέδριο, οι καλά σχεδιασμένοι κανόνε και διατάξει πρέπει να είναι σαφεί όσον αφορά την ερμηνεία και απλή στην εφαρμογή, μειώνοντα τον κίνδυνο σφαλμάτων και παρέχοντα δυνατότητα <clears throat> καθιέρωση απλουστευμένων μηχανισμών ελέγχου με βελτιστοποίηση σχέσης κόστους-οφέλους, κόστου αποτελεσματικότητα. Παράδειγμα των σοβαρών προσπαθειών που καταβλήθηκαν για την απλούστευση των καθεστώτων δαπανών αποτελεί η γεωργία. Ο κύριο τομέα τον οποίο το συνέδριο διαπίστωσε βελτίωση. Ωστόσο, η απλούστευση πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή. Η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιβάλλεται για την απλούστευση των κανόνων, η προσοχή μετά κατά την απλούστευση των κανόνων επιλεξιμότητα προκειμένου να αποφεύγεται η μείωση τη στοιχειοθέτηση των δαπανών. Επίση, φυστάται η προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι απλουστεύσει των προποθέσεων πληρωμών, οι οποίε στοχεύουν πρωταρχικά στη μείωση του διοικητικού φόρτου, του κόστου για του δικαιούχου ή των καθυστερήσεων δεν θα οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη αύξηση του κινδύνου πραγματοποίηση παράτυπων πληρωμών. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει αύξηση κινδύνου κατάχρηση κονδυλίων ή παρέκκληση χρήση και πρέπει να είμαστε στα συστήματα εποπτείας και ελέγχου αποτελεσματικοί. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας, ολοκλήρωσα την παρουσίαση των βασικών μηνυμάτων της ετήσιας έκθεσής μας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον, την εκτέλεση του προπολογισμού του οικονομικού έτους 2008. Η ετήσια έκθεση αποτελεί βεβαίω βασικό προϊόν του Συνεδρίου. Όπως όμως γνωρίζει η Επιτροπή σας δεν είναι το μοναδικό μέσο. Στην τρέχουσα εβδομάδα το Συνέδριο θα δημοσιεύσει επίσης ειδικές αιτήσει εκθέσεις για τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μετά την τελευταία διαδικασία χωρίς απαλλαγή στο συνέδριο ήδη κατήρθησε 15 ειδικέ εκθέσει σε σχέση με τα θέματα που κυμαίνονται από την επισητιστική βοήθεια μέχρι και ε, ε, για του απόρου ω και την ταμιακή διαχείριση τη Ένωση. Στι εν λόγω εκθέσει αφενό επισημένονται οι προκλήσει για τη βελτίωση τη δημοσιονομική διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερβαίνουν το στόχο τη περαιτέρω μείωση ε, των επιπέδων παράτυπων πληρωμών. Για να σα δώσω τα δύο πιο πρόσφατα παραδείγματα σε σχέση με την η ειδική έκθεση του συνεδρίου σε σχέση με τα μέσα διαχείριση αγορά στο τομέα του γάλακτο γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, επισημαίνεται ότι τα μέσα πολιτική σε ορισμένε περιπτώσει δεν επαρκούν για την επίτευξη των ευραίων και μάλλον αντικρουόμενων στόχων πολιτική που έχουν τεθεί. Ενώ η έκθεση και τα δίκτυα αριστεία και τα ολοκληρωμένα έργα στην κοινοτική πολιτική έρευνα υποδεικνύουν ότι τα προβλήματα που ε, αναφύονται και προκύπτουν όταν ένα πρόγραμμα δαπανών δεν διαθέτει σαφή λογική παρέμβαση ή ε, δείκτες επιδόσεων. Έτσι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώνει τη δέουσα προσοχή στα μηνύματα που διατυπώνει το ελεγκτικό συνέδριο στι αιτήσει και ειδικέ εκθέσει του κατά τη διαδικασία κατάτηση των προτάσεών τη για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την αναμόρφωση του προπολογισμού. Προ τον σκοπό αυτό το συνέδριο προτίθεται να καταρτήσει ένα δημόσιο έγγραφο που θα συγκεφαλαιώνει τα κύρια μηνύματα των, πρόσφατων εκθέσεών του και θα συμβάλλει περαιτέρω την παροχή συνδρομή προ την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο <clears throat> στο πλαίσιο των προσπαθειών για βελτίωση τη δημοσιονομική διαχείριση. Το έγγραφο αυτό θα επισημαίνει του τομεί ε, στου οποίου το συνέδριο διαπίστωσε ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ε, μείωση των παρατυπιών και βελτίωση τη δημοσιονομική διαχείριση. Η συνθήκη τη Λισαβόνα επίση ε, παρέχει και συνεπάγεται μεταβολέ στην λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε θα επηρεάζουν του αντίστοιχου ρόλου και αρμοδιότητε τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Αυτέ οι αλλαγέ θα έχουν Σημαντικέ επιπτώσει για το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου και αναμένεται ότι θα χρησιμεύσουν στην ενίσχυση των υποχρεώσεων λογοδοσία και στην αύξηση τη διαφάνεια, συμβάλλοντα κατά αυτόν τον τρόπο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η παρούσα χρονική στιγμή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανανέωση και μεταρρυθμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόσφατε ευρωεκλογέ μα έδωσαν ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο με ένα νέο πρόεδρο. Μετά από την ανανέωση τη εντολή τη θητεία του κυρίου Μπαρόζο, ω Προέδρου τη Επιτροπή και μια νέα Επιτροπή πρόκειται σύντομα να συνταχθεί, να καταρτιστεί. Ωστόσο, η σε περίοδου ανανέωση και μεταρρυθμίσεων είναι σημαντικό να αντλούμε διδάγματα από το παρελθόν Θεωρώ ότι το συνέδριο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο, καταρτίζοντα εκθέσει και διατυπώνοντα γνώμε, μέσω των οποίων όχι μόνο εντοπίζονται τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά και διατυπώνονται συστάσει. Γι' αυτό προσβλέπει το Συμβούλιο ιδιαίτερα στη συνέχιση τη συνεργασία του με τα άλλα εταιρικά θεσμικά όργανα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο τις παρούσες ευκαιρίες ε, για περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Eh, σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την ε, ενδελεχή σας παρουσίαση που αναφέρθηκε στην τις εργασίες που κάνατε τον περασμένο χρόνο. Πριν να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Κάλλας, θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πτυχές, κάποιες πτυχές που μου φάνηκαν πολύ σημαντικές και που προέκυψαν και από τη δική σας παρουσίαση. Καταρχήν, που πιστεύω ότι θα τη συμφωνείτε όλοι, δηλαδή συνολική απλοποίηση του νομικού πλαισίου. Οι κανόνες είναι πιο αποτελεσματικοί όσο πιο απλή είναι και αρκούν λίγοι κανόνες ώστε ε, από τη στιγμή που είναι σαφής και ευστηρία ακριβώς όσον αφορά το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας. μια άλλη πτυχή που νομίζω πως προκύπτει από την έκθεση και νομίζω πως αυτό είναι Σαφέ και από τα όσα είπε η Κομισιόν, θα πρέπει να γίνονται εποπτείες και έλεγχοι όχι μόνο από τα κρατημέλη αλλά και από την Κομισιόν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική η δραστηριότητα του ελέγχου η οποία να επιβαρύνει όλα τα, αυτά τα όργανα. Τώρα όσον αφορά τους ε, σκιές τις οποίες εσείς μας ε, περιγράψατε ε, σύντομα, νομίζω πως αφορούν την συμπεριφορά κάποιων κρατών μελών και ιδιαίτερα για πολύ λεπτά ζητήματα όπως αυτά των πολιετών διευθυντικών ταμείων ταμείων, καθώ και άλλη μια πτυχή που εσεί υπογραμμίσατε και σήμερα, δηλαδή την παραβίαση ή, εν πάση περιπτώσει, την μη τήρηση του κανόνα για του μεδοτικού διαγωνισμού. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσέξει η Κομισιόν γιατί πέρα από τα σφάλματα, τα σημαντικά σφάλματα τα οποία υπογραμμίζει το ελεγκτικό συνέδριο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μπορεί να υπάρχουν και πολύ πιο σοβαρές υποθέσεις όπως όλοι γνωρίζουμε που είναι οι απάτε και οι παρατυπίες που είναι οι ε, ε, ε, πιο επικίνδυνες. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Κάλλας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Σίλβα Καλντέιρα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για την ε, τελευταία αυτή ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στα πλαίσια της Κομισιόν Μπαρόσο και θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί πρόκειται για την καλύτερη ετήσια έκθεση που είχαμε μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν παρουσιάστηκαν οι συστάσεις και τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου με τόσο ξεκάθαρο και επικοδοματικό τρόπο. Και βλέπω το διάλογο και η συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο δεν ήταν τόσο επιτυχη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καλντέιρα και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για την καλύτερη δυνατή έκθεση που είχαμε και από μία άλλη βέβαια προσέγγιση, από μία άλλη οπτική γωνία. Βλέπετε στη γραφική αυτή παράσταση πώς έχουν εξελιχθεί οι εργασίες του λεπτικού Συνεδρίου από το 1994 και μετά. Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα και στην έκθεση του κυρίου Καλντέιρα και όπως βλέπετε τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται και από το 2004 και μετά το κόκκινο αυτό τμήμα έχει μειωθεί κατά το ίμιση. Για πρώτη φορά η γεωργία αντιμετωπίζεται στο σύνολό της και η ε, ομάδα πολιτικής εκπαίδευση και ε, ιδιότητα του πολίτη εμφανίστηκε και αυτή με πράσινο χρώμα φέτος και βελτιώνονται τα αποτελέσματα. Όσον αφορά την ε, κόκκινη ε, περιοχή, την κόκκινη ζώνη, αυτή αφορά μόνο το 30% της περιοχής συνοχής. Μόνο εκεί πέρα δεν εντυπίστηκε κάποια πρόοδος. Ήταν αμενόμενο όμως αυτό για το 2008 το λεκτικό συνέδριο δεν έλεγξε τους, τις πληρωμές που γίνανε στα πλαίσια των νέων συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για, το, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Συνολικά, έχοντας ακούσει την παρουσίαση του Προέδρου σήμερα το πρωί, σημειώνω το ελεγκτικό συνέδριο δίνει μια ξεκάθαρη γνωμοδότηση για τους λογαριασμού και ότι το 2008 είναι το καλύτερο δυνατό έτος που είχαμε μέχρι στιγμής όσον αφορά τα οικονομικά της Ένεσης. Η έκθεση αυτή μας ε, δείχνει βέβαια ότι πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συζητήσει περισσότερο τις ε, διορθωτικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια δικασία απαλλαγή και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής σας και με τον εισηγητή κύριο Λιμπεράτσκι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, παρατηρήσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί και ξέρω ότι και εγώ ίδιος αλλά και οι συναδελφοί μου στο μέλλον θα εργαστούμε πολύ για τις ακροάσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της απαλλαγής για το προπολογισμό που θα γίνουν στις 2 Δεκεμβρίου. Εγώ θα έρθω στις 26 Ιανουαρίου πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των ακροάσεων αυτό και θα έχουμε τότε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες του προπολογισμού στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Χαίρομαι όμω πάρα πολύ που μα δίνεται ήδη σήμερα μια πρώτη ευκαιρία για να μιλήσουμε περισσότερο για την αύξηση του ελέγχου και τη εποπτεία, για την αύξηση τη απλούστευση των λογαριασμών. Και αγαπητά μέλη τη Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αποφαθώ για τα σημεία αυτά. Αναφερθήκαμε επίσης στο ζήτημα του ε, shared management, της ε, κοινή διαχείρισης, της ε, συνδιαχείρισης. Αναφερθήκαμε στο ζήτημα αυτό από την οπτική γωνία της ανάκτησης, της ευθύνης για τους και πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι από την αρχή τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια είδαμε μια συνεχή αύξηση και βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Και έχουμε και ξεκάθαρα παραδείγματα. Οι πληροφορίες πλέον είναι πιο πλήρεις, είναι καλύτερες και εξ αρχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τώρα στις εκθέσεις, ε, τις εκθέσεις δραστηριοτήτων βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται πλέον ε, νέα μέσα όπως ε, η ε, προσωρινή πάυση κάποιων πληρωμών που ισχύουν για κάποια κράτη-μέλη και για το ζήτημα αυτό δεν αντέδρασαν θετικά ορισμένα κράτη-μέλη αλλά ακόμα και κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή και ένα πράγμα που πρέπει να τονίσω είναι ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Επιτροπών των Αρμοδίων για τον Προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα πάρα πολύ καλή και η συνεργασία αυτή μας ε, επέτρεψε να έχουμε μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και μια καλύτερη ανάλυση των αιτήσεων εκθέσεων που υποβάλλουν ε, τα κράτη-μέλη και των αιτήσεων αυτών περιλήψεων που χρησιμοποιούμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συζητήσουμε περισσότερο λεπτομέρειες αυτές και στο μέλλον, κατά τη διάρκεια των ε, ακροάσεων που θα γίνουν για την απαλλαγή από τον προπολογισμό. Σήμερα συζητάμε τη γενική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Κάλλας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το επαληθεύσαμε και από την ανάλυση ανάμεσα στο παρελθόν και το πρόσφατο παρελθόν ότι υπήρξαν πολύ σημαντικές βελτιώσει που επιτεύχθησαν χάρη στην δουλειά τη Κομισιόν. Νομίζω πως είναι σημαντικό να βρεθεί μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων που μας προτείνει η δημόσια χρηματοδότηση και τις ε, ακραίες ε, τυπικότητες. Δηλαδή κάποιες φορές η υπερβολική γραφειοκρατία και ε, τυπικότητα μπορεί να μας εμποδίσει από το να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και κάτι ακόμα που νομίζω προκύπτει από την έκθεση του, του Ελεκτρικού Συνεδρίου είναι ότι υπάρχει προφανή ε, διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα κράτη-μέλη υπάρχουν που σέβονται συγκεκριμένα όλου τους κανόνες και όλες τις υποδείξει, ενώ άλλα χρησιμοποιούν τις δικές τους συνήθειες και πάντα είναι στα κόκκινα. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ώστε οι κανόνες να είναι οι ίδιοι για όλους και να εφαρμόζονται από όλου. Ο κύριος Λιμπεράτσκι που είναι ο εισηγητή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επίτροπή, κύριε Επίτροπε Κάλλας. Εδώ και κάποια χρόνια έχω την χαρά να ακούω τις εισηγήσεις σας στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής και σήμερα η παρουσίασή σας δείχνει πως έχετε λόγος να είστε χαρούμενος. Και ναι, οι εκθέσεις παρουσιάζονται είναι καλύτερες χρόνο με το χρόνο. Έχουμε καλύτερη εικόνα για τη βελτίωση και τη σωστή διαχείριση των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη. Όταν θα αναφερθώ στην έκθεση του, Συμβου... του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην έκθεση του κυρίου Καλντέρα. Η έκθεση αυτή, και πιστεύω πως θα συμφωνείτε με, μαζί μου, θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής. Αυτή η γενική τάση που ε, οδεύει προς μια βελτίωση σηματοδοτείται ωστόσο από ελλείψεις που ακόμα και σήμερα επιμένουν και παραμένουν στους ίδιους τομείς. Τρεις είναι οι εν λόγω τομείς. Τρεις τομείς που δημιουργούν πρόβλημα και που γενικά λεκιάζουν αυτήν την ε, θετική τάση. Ταμείο Συνοχής και Διευθυντικά Ταμεία, εξωτερικές δράσεις της Κομισιόν και τέλος και αυτό ίσως να χρησιμοποιούμε διαφορετικά κριτήρια, όμως υπάρχει αυτό το χάσμα ανάμεσα στα κατημέλη, το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Επιστήνω την προσοχή σας σε αυτό που βλέπουμε στην ε, σελίδα 136 της έκθεσης. Εδώ αξιολογείται το σύστημα εποπτείας και ελέγχου σε έναν μόνο τομέα στα κρατη Σε αυτό το τομέα έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης. Υπάρχουν πληροφορίες για τις διορθώσεις που έχει επιφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν 10 τομείς όπου οι πληροφορίες δεν είναι ικανοποιητικές ή είναι μερικώς ικανοποιητικές. Άρα λοιπόν από τους 16 τομείς μόνο 6 τομείς είναι αυτοί όπου δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία τους. Δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις εργασίες είναι η καταγραφή των διορθώσεων, η διόρθωση των σφαλμάτων και η δήλωση των προβλημάτων στην Όλαφ. Εγώ πιστεύω πως υπάρχει κάποια αντίσταση για διάφορους ε, τομείς και εδώ θα πρέπει να ε, εστιάσουμε την προσοχή. Διαστοτικά ταμεία και ταμείο συνοχής. Από την άποψη της Κομισιόν είναι πολύ αρνητικό να βλέπουμε εδώ το ποσοστό σφάλματος πάνω από 11% δηλαδή το ίδιο με πέρσι και με δύο χρόνια πριν και Πέρσι γίνανε οι ίδιες συζητήσεις στο πλαίσιο αυτής της ε, Κομισιόν που διερωτηθήκαμε αν έπρεπε να δοθεί απαλλαγή για αυτό το κομμάτι του προπολογισμού ή όχι. Στη συνέχεια είχαμε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε 21 σημεία όπου έπρεπε να υποδείξουμε πώς από τα κονδύλια από τα έτη 2000 μέχρι 2006 θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάκτησης και απάντηση ήταν ότι πολύ λίγα από αυτά θα ανακτώνταν. Έπειτα, πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα του 2007. Η απάντηση είναι δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε πώς να διορθώσουμε αυτά τα σφάλματα και Τρίτον, πώς θα ελαχιστοποιήσουμε με ριζικό τρόπο το ποσοστό σφάλματος για το 2008 και 2009 και αυτή η ελαχιστοποίηση, η μείωση για το 2008 δεν υπάρχει, γιατί το ποσοστό σφάλματος εξακολουθεί να είναι παραπάνω από το 11%. Ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι να σκεφτεί με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να σκεφτούμε τον καταμερισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο των διαφόρων ε, θεσμών που είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Κύριε Καλντέρα, εσείς αναφέρετε κάποιους τομείς. Μη τήρηση των κριτηρίων από τα διάφορα προγράμματα, προγράμματα που που υπάρχει κακοδιαχείριση, κακή και η συμπεριφορά των κρατών μελών. Η κατάσταση έχει ως εξή. Ανάμεσα στο 2000 και το 2006 ολοκληρώνονται διάφορα προγράμματα και για το 2007, ε, την περίοδο μάλλον 2007 μέχρι 2013, βρισκόμαστε στο 40% της αλλά αυτό δεν το βλέπουμε στην πράξη σε σχέση με τους ε, δικαιούχους. Δεν είναι αντικείμενο βέβαια αυτό της σημερινής μας συνεδρίασης, αλλά Πιστεύω πως ρόλος μας είναι να συνειδητοποιήσουμε το τι θα μπορούσε να συμβεί. Ε, γινόμαστε ίσως μάρτυρες ε, ενός σημαντικού γεγονότος αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για αυτή τη σώρευση την οποία ανέφερα ήδη. Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει σώρευση σφαλμάτων. Και αυτό γιατί, γιατί ε, τα κράτη-μέλη συχνά ε, θεωρούν πως οι καταβολές για την περίοδο 2007-2013 ε, είναι έσοδα στον προπολογισμό τους και τα κονδύλια αυτά δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε για τους στόχους για τους οποίους έχουν εκταμιευθεί. Στη συνέχεια αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τη λειτουργία των ε, ταμείων. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν διαπιστώνω πως υπάρχει βελτίωση σε κάποιους τομείς για τους οποίους είχαμε ανησυχίες, ε, δηλαδή έρευνα, ενέργεια, μεταφορές. Και εδώ προσεγγίζουμε αυτό που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε αποδεκτό. Εξωτερικές δράσεις τώρα, δεύτερος ε, μεγάλος τομέας που από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι για το Ταμείο Συνοχής και τα Διευθυντικά Ταμεία. Ε, το ποσοστό σφάλματος πέρασε από το 50% στο 31-32%. Αυτό είναι βέβαια βελτίωση της τάξης του 40%. Όμως ε, το ποσοστό σφάλματος παραμένει εξαιρετικά υψηλό πολύ πιο υψηλό από αυτό που έχουμε για το Ταμείο Συνοχής και τα Διευθυντικά Ταμεία. Ο κύριος Καλδέρα μας πρότεινε να συνεχιστεί η απλοποίηση των κειμένων και των διαδικασιών. Εγώ επιστήνω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε ναι στην απλοποίηση εις βάρος της διαφάνειας. Και εδώ, αν κοιτάξουμε το γράφημα που μας ε, δείχνετε, τα κόκκινα τμήματα βλέπω το 1994 και διαπιστώνω πως η διαφάνεια είναι ε, ε, σημαντική όσον αφορά την παραλαβή των, χρημα... των κονδυλίων. Και εγώ θεωρώ πως και, και, και εδώ σας απευθύνω ερώτηση κύριε Κάλλας. Η Κομισιόν θεωρεί πως είναι αρκετά ισχυρή σε σχέση με τα κράτη-μέλη. θεωρεί ότι είναι καταλήλως εξοπλισμένη απέναντι στο Συμβούλιο ώστε να καλύψει αυτές τις ελλείψεις και επιτέλους να λάβει τις αποφάσεις που θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες και κατά δική μας άποψη. Αν η απάντησή σας είναι ναι, θα ήθελα να γνωρίζω πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε. Ευχαριστώ το Ευρωβουλευτικό Συνέδριο και ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χάτζη Μαρκάκη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν κύριε Καλτέρα θα ήθελα να σας συγχαρώ ειλικρινά για την εξαιρετική σας παρουσίαση καθώς και για αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα αριθμό. Κύριε Σίμων Κάλλας, σας ευχαριστώ γιατί μας δείξατε αυτό το γράφημα, γιατί πολλές φορές μια εικόνα δείχνει περισσότερα από ό,τι χίλιες λέξεις και ο κύριος Καλντέρα και κύριε Καλντέρα και κύριε Κάλλας ε, θέλω να σας συγχαρώ και για την καλή συνεργασία σας. Όμως υπάρχουν ε, ακόμα τομείς ε, όπου τα πράγματα είναι πιο αρνητικά. Χαιρόμαστε για τις πράσινες γραμμές, χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι εκεί όπου υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί είναι αποτελεσματικοί, όπως για παράδειγμα για τη Γεωργία έχουμε το σύστημα Ajax, το οποίο θα πρέπει σωστά να επενεθεί και εδώ βλέπουμε πως ε, έχουμε ε, πολλές βελτιώσεις, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί και με την εντολή ε, του κυρίου Κάλλας και του κυρίου Μπαρόζο και ελπίζω πως η Κομισιόν Μπαρόζο 2 θα επιτρέψει την περαιτέρω βελτίωση των πραγμάτων. Ωστόσο βλέπουμε που υπάρχουν, ξεκολουθούν να υπάρχουν σκιές. Υπάρχουν σκιές εκεί όπου τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, στη διάθεσή τους κοινοτικού μηχανισμούς. Εκεί όπου τα κράτη-μέλη είναι αμελή και δεν δίνουν την κατάλληλη προσοχή. Και όταν μιλάμε για 11% κύριε Καλντέρα, ε, είναι 4 δις ευρώ δις ευρώ των φορολογούμενων που εξαφανίζονται ή που εν πάση περιπτώσει καταβάλλονται με παράνομο τρόπο, παράτυπο τρόπο. Οπότε είναι αποτυχία, ναι, των κρατών μελών, αυτό είναι σαφέ. Εδώ εμείς μπορούμε να συγχεζόμαστε να θυμώνουμε, να τους ε, δακτυλοδείχνουμε, αλλά αυτό που εμένα με ανησυχεί και θα ήθελα να δω και να σας ρωτήσω, όπω και ο κύριος Λιμπεράσχη, μήπως είναι δυνατόν από πλευρά της Κομισιόν να επιμείνουμε περισσότερο στα κράτη-μέλη, ε, να τους πιέσουμε περισσότερο. Δεν υπάρχει άλλη λύση κατά την άποψή μου. Είναι χρήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αλλά ε, για το ευρύ κοινό αυτά τα χρήματα θεωρούνται χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστεύουν οι πολίτες και θα έπρεπε να είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι απέναντι στα κράτη-μέλη που επανειλημμένως και μάλιστα υπάρχουν διάφοροι ύποπτοι που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε λογαριασμό από αυτά τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν να είναι πιο αυστηρή. Ε, ε, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να σας βοηθήσει. υπάρχει μεγάλη πίεση και χάρη σε αυτή την πίεση έχουμε και καλύτερη συνεργασία μεταξύ μας. Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί. Να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρο για αυτό του έξι τομείς κλειδιά και νομίζω πως είναι πολύ θετικό που είχατε το θάρρος να πάρετε θέση για αυτές τις διάφορες πολιτικές. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει μόνο η συνοχή. μα είπατε ότι για παράδειγμα στα θέματα έρευνα υπήρχαν σφάλματα και μάλιστα εδώ εσείς ε, το συνδέετε με την, ε, τον περίπλοκο χαρακτήρα. Και έπειτα υπάρχει τώρα μία ακρόαση που αφορά ακριβώς τη μείωση της γραφειοκρατίας σε θέματα προγραμμάτων πλαισίου και προσπαθούμε πραγματικά να μειώσουμε την ε, ε, περιπλοκότητα αυτή, αλλά έχετε δίκιο όταν μας λέτε πως χρειάζεται απλοποίηση της εφαρμογής. Και ως προς αυτό νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Ε, δεν πρόκειται για την ίδια τον έλεγχο, πρόκειται για τους κανόνες του εφαρμοστικούς που θα πρέπει να απλοποιηθούν. Και εδώ είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόταση από πλευρά σας. Και τέλος να ευχαριστήσω άλλη μια φορά, να συγχαρώ μάλλον το ελεγκτικό συνέδριο για την εξαιρετική της εργασία. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου έχει βελτιωθεί πολύ. Είναι πιο ευανάγνωστη αυτή τη στιγμή, πιο σαφής. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον Επίτροπο προσωπικά, καθώς επίσης και όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάρτιση της έκθεσης αυτής. Έχουμε επίσης και πίνακες με σαφή αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι έχουν υποβληθεί πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, οι οποίες απέδωσαν καρπούς. Πρόκειται λοιπόν για επιτυχία τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πολύ σημαντική επιτυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν πηγιάδικα λοιπόν όλη η σκληρή δουλειά που έλαβε χώρα και είδαμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια μπορεί να μην γίνανε όλες οι αλλαγές που θα θέλαμε να είχαν γίνει ή να μην είχαν γίνει τόσο γρήγορα. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να εξασκούμε πίεση προκειμένου να σημειώσουμε και νέες επιτυχίες στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να θαρρύνω τους ευρωσκεπτικιστές συναδέλφους να είναι πιο δίκαιοι. Ξέρω ότι η δήλωση εξοπιστίας δεν είχε δοθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι ε, εξοικειωμένα ακόμα με την ε, δημοσιονομική διαδικασία της δήλωσης αξιοπιστίας να επικεντρωθούν σε αυτήν περισσότερο. Το μήνυμα το οποίο περνάει μέσω της δήλωσης αξιοπιστίας είναι ένα μήνυμα επιτυχίας και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ε, επιμείνουμε στα θετικά σημεία της έκθεσης προτού περάσουμε στα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Να δούμε που οι προσπάθειές μας δεν έχουν αποδώσει καρπούς ακόμα και στους τομείς εκείνους να επιμείνουμε. Σε τι συμπέρασμα λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε βάσει των κειμένων αυτών. Πολλοί έλεγχοι έχουν γίνει, αυτό το βλέπουμε. Και όσοι έλαβαν τελικά πληρωμές θεωρούν πολλές φορές ότι ε, ο έλεγχος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ήταν ε, υπερβολικός. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε περισσότερο για το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι και να καταλήγουν στα σωστά αποτελέσματα, σωστά πορίσματα. Όταν μιλάμε για ανάκτηση, το πρόβλημά μας δεν είναι η ανάκτηση αυτή καθ' αυτή. Ουσιαστικά θέλουμε να βελτιώσουμε το όλο σύστημα προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα με την ανάκτηση. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ζητήματα αυτά τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υπογραμμίσει με κόκκινο χρώμα στον ε, πίνακα των αποτελεσμάτων. Ακούγοντα και τον κύριο Χατσιμαρκάκη, πιστεύω και εγώ ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στο όλο σύστημα, αλλά υπάρχουν και αρνητικά όσον αφορά την ανάλυση του κινδύνου. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στην ε, γεωργία, και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό το 2% της αξιοπιστίας για την γεωργία θα πρέπει να το δούμε και αυτό σαν μια επιτυχία, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες, ε, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που έχουν φτάσει το 12 ή το 13%, ενώ ε, ο αντίστοιχο, το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες όπως η Γερμανία είναι πολύ μικρότερο. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμη μια πολύ μεγάλη απόκληση όσον αφορά τα ποσοστά αξιοπιστίας για συγκεκριμένου τομεί πολιτική. Μιλώντας τώρα για συγκεκριμένες επισκέψεις αποστολές, π.χ. στη Ρουμανία, θα πρέπει αυτές να γίνουν και να δούμε τελικά τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν ε, εντοπιστεί ε, προβλήματα. Θα πρέπει ενδεχομένως να ε, ενεργοποιηθούν και συγκεκριμένε γενικές διευθύνσει και επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να επιτύχουμε ακόμα κάποιες σημαντικές βελτιώσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φτάνει στο τέλος της θητείας της, αλλά και με την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβουμε δράση στο μίσο που απαιτείται κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τομείς αυτοί όπου έχει εντοπιστεί μια κάποια χαλάρωση. Γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς ακόμα τι έχει γίνει με τους πόρους, με τα κονδύλια σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να φτάσουμε, να είμαστε δηλαδή σίγουροι ότι τα κονδύλια δαπανούνται βάσει της πολιτικής που έχει εγκριθεί Αυτό το έχουμε πετύχει σε κάποιους τομείς και αυτό αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία. Ξέρω ότι πρέπει να γίνει ακόμα πολύ σημαντική δουλειά στο μέλλον, είμαι όμως πολύ αισιόδοξο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Πρόεδρό του Καλντέιρα για την σημαντική δουλειά που έχουν κάνει και να τον ευχαριστήσω επίσης και για όλα τα έγγραφα τα οποία μας έδωσε. Στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών Ήρθατε σήμερα και μιλήσατε και μας είπατε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτό μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε και εμείς σε ποιο βαθμό η δικιά μας εργασία έχει οδηγήσει σε κάποια θετικά συμπεράσματα, σε κάποιες επιτυχίες. Είναι πολύ σημαντικό επίση να γνωρίζουμε πού θα πρέπει να επισέλθουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε, σε ποια προβλήματα θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Από τη μια μα λέτε ότι χρειαζόμαστε καλύτερα συστήματα εποπτεία και ελέγχου και από την άλλη μα λέτε ότι χρειάζεται και μια πλούστευση ε, του νομικού καθεστώτο. Αυτό εκ πρώτη όψη μπορεί να φαίνεται κάπω αδύνατο όσον αφορά την βελτίωση των συστημάτων ε, ελέγχου και εποπτείας. Ενδεχομένως εδώ πέρα να θέλετε πιο εντελεχείς ελέγχους αλλά ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο γραφειοκρατίας και μα λέτε επίση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα του διαθέσιμου πόρου και να οδηγούμεθα σε λιγότερα σφάλματα. Απαιτείται επίση, είπατε, καλύτερη διαφάνεια για το πώ δαπανούνται τα χρήματα και το πού δαπανούνται τα χρήματα. Σαφώ εμεί ω Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημεία αυτά και αν καταφέρουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, τότε αυτό θα ήταν και το ιδανικό σίγουρα. Πρέπει επίση να γνωρίζουμε σε ποιου τομεί τα πράγματα λειτουργούν θετικά. Στα πλαίσια τη ε, Επιτροπής μας και με τη βοήθεια των κρατών μελών θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Και να δούμε και το θέμα των ετούντων σε σχέση με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι ανταλλαγές μαθητών, είτε είναι θέματα έρευνας, είτε είναι διαθροτικά ταμεία και κονδύλια διαθροτικών ταμείων. Μιλώντας με τους ετούντες πάντα ακούω την, το παράπονο ή την κατηγορία ότι τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι όγκου τηλεφωνικού καταλόγου τα έντυπα αυτά. Και για παράδειγμα δάσκαλοι, καθηγητές που για το σχολείο τους ζητούν τέτοια μέτρα δεν έχουν την τόλμη να θέσουν τέτοιες αιτήσει, διότι θα χρειαζόταν φοροτεχνικός ή νομοτεχνικός για να τα συμπληρώσουν. Πώς μπορούμε να πετύχουμε την απλούστευση λοιπόν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ας το πω έτσι, τα ωφελήματα, τα προτερήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες να καταστούν σαφέστερα με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι πιο προσπελάσιμα, με, ευκολότερη πρόσβαση, με διασφάλιση διαφάνειας και με τους ελέγχους που θα διατηρούνται σε ένα τέτοιο μέτρο που θα αποκλείονται τα λάθη και τα σφάλματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει βέβαια άμεσα, αλλά ακούγεται σαν τετραγωνισμός του κύκλου ένα τέτοιο όνειρο, ως χήμερα ασχολούμαι αυτό το θέμα σε ένα μικρότερο εύρος προγράμματος από πλευρά σχολείων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά ε, ήταν ε, το, ε, η δομή των δικών μας ομοσπονδιακών δομών και αυτό είναι μια επίκριση που μπορεί να εισακουστεί. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης για αυτά τα προγράμματα είναι τόσο υψηλή ώστε το κόστος, οι συνολικές δαπάνες είναι συντριπτικές. Το πρόγραμμα, τα κονδύλια που δίνει αυτό το πρόγραμμα για την, την κάτω Σαξονία αντισταθμίζονται από τις δαπάνες. Δηλαδή τα όσα είναι όφελος ως καθαρή φορά αντισταθμίζονται από τις δαπάνες που μας προκαλούνται και έτσι προκαλούνται σκέψεις σε ένα ελεγκτή, δημοσιονομικό ελεγκτή. Αν πρώτον είναι σωστό κάτι τέτοιο, διότι θα ήταν πολύ αρνητικό κάτι τέτοιο, αν μηδενικό ποσό είναι αυτό το οποίο δαπανάτε για παράδειγμα, ή αν ένα προσχηματικό στοιχείο ως λόγος είναι για παράδειγμα η εξοικονόμηση συμπληρωματικών κονδυλίων. Θα λόγο αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρέσλε και ο κύριο Χατζημαρκάκης. Στο μέλλον να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη αυτά τα κονδύλια και τι κάνουν από πλευρά του, Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα για το πώς οι έλεγχοι υλοποιούνται και πώς οι έλεγχοι διαμορφώνονται και πόσο συνεργάζονται τα κράτη-μέλη και τι γίνεται με τις δυνατότητες αυτές όπου τα κονδύλια για παράδειγμα με κακό τρόπο διαχειρίζονται. Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που είπε ο κύριος Κάλλας ότι μια τέτοια προσέγγιση από τα κράτη-μέλη δεν θα ε, προκαλούσε μεγάλη ικανοποίηση. Αυτό άμεσα το πιστεύω. Όμως ως Ευρωβουλευτής θα έλεγα, όμως προκαλεί ενθουσιασμό από πλευράς πολιτών που μας εξέλεξαν να κάνουμε τη δουλειά μας ως Ευρωβουλευτές. Και αν έχουμε σαφή επιχειρήματα στις επόμενες ευρωεκλογές ότι συγκεκριμένα προβλήματα σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη έγκυνται σε συγκεκριμένα προγράμματα και αν έχουμε μια σαφή ημερήσια διάταξη από κοινού με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο χρόνος που έχουμε να εργαστούμε για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, όμως να πούμε με σαφή τρόπο πού βρίσκονται οι ευθύνε. Τότε εξυπηρετούμε σωστά την Ευρώπη, πιστεύω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στάρης. Ευχαριστώ πολύ και εγώ Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, ιδιαίτερα φυσικά τον πρόεδρο κύριο Καλντέρα για τον τρόπο που εργάστηκαν, το θετικό έργο που επετέλεσαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και ιδιαίτερα για εφέτο για τι ειδικέ εκθέσει, που είναι ενδιαφέρουσε εκθέσει. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάλλα, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, για την παρέμβασή του. Και από το γράφημα βλέπω ιδιαίτερα ότι η κατάσταση μεταξύ 94 και 99 ήταν ιδιαίτερα αρνητική, ιδιαίτερα δεινή. Ήταν η περίοδο που εδώ στην Ευρωβουλή και στην Επιτροπή Ελέγχου για τον προϋπολογισμό στην Ευρωβουλή κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να κινητοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να λάβει μέτρα. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια στην πτώση της Επιτροπής Σαντέρ και αυτό το οποίο έκανε το Κοινοβούλιο από το 1999 μέχρι σήμερα και οδηγηθήκαμε σε βελτιώσεις και είναι σημαντική υπόθεση αυτή. Η συνεισφορά της Ευρωβουλής και η πίεση που άσκησε η Ευρωβουλή από το 1999 έως το 2009, 10 ολόκληρα χρόνια, δεν πρέπει να υποτιμάται. Ο κύριος Καλτέρα στις 11 και 4 πρέπει να αποχωρήσει και θα είμαι εν συντομία θα τοποθετηθώ. Διάβασα την έκθεση και μία από τις κυριότερες παραγράφους όσον αφορά τον τύπο και την ε, ε, συνέντευξη τύπου και τα σχετικά με την τεκμηρίωση είναι σε σχέση με το 16 και 17 όπου αναφέρεται ότι στα ταμεία συνοχής, δηλαδή διαρθωτικά ταμεία, κοινωνικό ταμείο, αυτό το ευρύτερο ταμείο συνοχής, ότι εκεί 11% αχρεωστήτως κατεβλήθησαν ποσά πλεονάζοντα υπερβολικά ποσά. Θα θέλω ο κύριο ε, Κάλλα, αρμόδιο επίτροπο για την καταπολέμηση απατών και ο κύριο Καλντέρα, επικεφαλή του ελεγκτικού συνεδρίου, να, πει, να μας πούν αν είναι δυνατόν ακόμα με σαφέστερο τρόπο να διατυπωθεί αυτή η παράγραφο και να είναι ακόμα οξύτερη. Διότι σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και σχεδίων πληρώθηκαν υπερβολικά κονδύλια. 11% υπερβολικά πλεονάζον δυναμικό. Είναι ακριβώ κατά τα άλλα όπω και πέρυσι και πρόπεση 12% είχαμε τότε. Και τι γίνεται τώρα, σε ποιο ποσό έχει υπολογιστεί το 24,8 δις από, το από το... την υποσημείωση. 11 ε, είναι, 2,7 δις, όχι 4 δις που ανέφερε ο κ. Χατζημαρκάκης, 2,7 δις. Είναι το σωστό ποσό αυτό, είναι η σωστή ανάγνωση, η σωστή ερμηνεία αυτής της παραγράφου. Διότι κατά τα άλλα αύριο θα έχουμε δημοσιεύματα στον τύπο, στις εφημερίδες. Θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία οι εφημερίδες. Είναι η ορθή ανάγνωση αυτής της παραγράφου 11% υπερβολικές δαπάνες που καταβλήθηκαν από το συνολικό ποσό των 24,5 δις. Αυτά έχω να ρωτήσω. Έχω και πολλές άλλες ερωτήσεις, αλλά βρίσκεται ενρευστό εν εξελίξει η διαδικασία και έχω ευκαιρία και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριος Μπάτσεβης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, Πρόεδρε. Πράγματι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στις ε, παρατηρήσεις των συναδέφων για τις ευχαριστίες που εξέφρασαν προς το ελεγκτικό συνέδριο για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και να ευχαριστήσω για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην προπαρασκευή αυτών. Όμως η δική μας Επιτροπή Ελέγχου του Προπορισμού θα έπρεπε περισσότερο να επικεντρώνεται στα στοιχεία όπου υπάρχουν τα προβλήματα, στους τομείς των προβλημάτων. Πρώτον και κύρια, στο Ταμείο Συνοχής. Δεύτερον, στις μεταφορές και στον τομέα των ερευνών. Και επιπλέον, στα σφάλματα που δια, ανοιχνεύονται και το ποσοστό σφαλμάτων. Όμως σήμερα θα έπρεπε να θυμηθούμε κάτι τι συνέβαινε στο παρελθόν. Η πλειοψηφία, η πλειοψηφία των νέων κρατών μελών εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 με τελείως διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις και τελείως διαφορετική πείρα και παρελθόν Τότε θεώρησαν τα νέα κράτη-μέλη ότι τα κονδύλια που δινόντουσαν από πλευρά του προπολογισμού τη Ένωση θα έπρεπε να εγγράφονται σε ένα διαφορετικό κονδύλιο, όπω επιπρόσθετα κονδύλια, και δεν θα έπρεπε να εντάσσονται και να συμπεριλαμβάνονται στον εθνικό προπολογισμό. Όμω στη συνέχεια υπάρχουν και κανόνε και διατάξει, τι πρέπει να κάνουμε και πώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα κονδύλια, αυτού τους πόρους, ποιε προτεραιότητε θα πρέπει να είναι σεβαστέ κτλ. Σήμερα τα νέα κράτη-μέλη ήδη δρούν και αντιδρούν σε ένα πολύ καλύτερο ε, σε πολύ καλύτερα βάθρα. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών, μάλιστα πρέπει να πω οπωσδήποτε συμφωνώ με τους συναδέφους μου που ανέφεραν ότι προσπαθούμε βέβαια να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και είναι χειμερικό αυτό το εγχείρημα. Διότι αφενός κάνουμε λόγο για την ανάγκη απλούστευσης. Από την άλλη όμως πλευρά γίνεται λόγος για καλύτερους ελέγχους και καλύτερη εποπτεία. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω και μια ερώτηση. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για όλο αυτό το εγχείρημα. Τα κράτη-μέλη τα ίδια σήμερα δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ στην απλούστευση των διαδικασιών, στην απλοποίησή τους. Διότι μέσω απλοποίησης θα ε, αντιμετώπιζαν αυξημένες ευθύνες, ε, αυξημένο επίπεδο ευθυνών. Από την άλλη πλευρά παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο όλα εξαρτώνται από την ικανότητα και η δυνατότητα κάθε εθνικής κυβέρνησης να απορροφά και να χρησιμοποιεί τα διατηθέμενα κονδύλια κονδύλια. Γι' αυτό ένα πράγμα είναι σαφέ. Θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε την κατάσταση ω έχει σήμερα, την ενισχύει κατάσταση και να αναθεωρήσουμε τι διαδικασίε και διεργασίε. Γνωρίζετε ότι πολλέ φορέ δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Έχω υπόψη την ερμηνεία, για παράδειγμα, των κανονισμών και κανόνων όσον αφορά του τους Ευρωπαίου υπαλλήλου, τα στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, να απλουστεύσει τις διαδικασίες και διεργασίες και να τοποθετήσει ταυτόχρονα υπευθύνους υπαλλήλους που θα είναι αρμόδιοι για την ερμηνεία του ενός ή άλλου θέματος κανονισμού και διατάξεων. Αυτό θα συνεισέφερε να αποφύγουμε στο μέλλον επικάλυψη προσπαθειών και λανθασμένες ερμηνείες. Θα είχαμε και μια καλύτερη κατανόηση ταυτόχρονα για την εφαρμογή των κανονισμών και κανόνων και θα αποφεύγαμε τον κίνδυνο να ηγερθεί η κατηγορία κατάχρησης ή κακής χρήσης των κονδυλίων από πλευράς μας. Ο κύριος Λιμπεράσκι σωστά ανέφερε την ανάγκη μιας, ενός καλύτερου συσχετισμού με μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων. Όταν θα αλλάξουν και αν αλλάξουν οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το βάθος και τη βάση με την οποία εργαζόντουσαν τα νέα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα. Επίσης θεωρώ ότι οι εκθέσεις που παρουσιάζονται στα, σε σχέση με τα κράτη-μέλη και από τις διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να απλουστεύονται και αυτές. Θα πρέπει να έχουμε απλουστευμένες εκθέσεις που θα αναφέρουν απλά ποσά, αριθμητικά μεγέθη, προβλήματα, σφάλματα και έτσι θα είμαστε σε θέση να είμαστε αποτελεσματικοί όπως αναμένουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανδρεάσεν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γιατί αν κάτι τελικά έχει βελτιωθεί πολύ σημαντικά, αυτό είναι η ποιότητα των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, σημειώνω το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται στους λογαριασμούς, λέγοντας ότι παρουσιάζουν μία αντιπροσωπευτική καλή εικόνα των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο όμως δεν χρησιμοποιείται όρο όρος true, ότι δίνει μια αληθινή εικόνα και χρησιμοποιείται μόνο ο όρος fair στα αγγλικά. Αν δείτε διάφορες παραγράφους που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία των λογαριασμών, γίνεται αναφορά σε αδυναμίες του συστήματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα των δημοσιονομικών πληροφοριών και να συγκεκριμένα στον τομέα της προχρηματοδότησης όπου έθεσα ένα ερώτημα προς τον ε, ε, Chief Accounting Officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να γνωρίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η αποψή της σε σχέση με, την, ε, με τα ποσά προχρηματοδότησης τα οποία έχουν προβλεφθεί όσον αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο οι προλαλήσαντες, γιατί τελικά, στη τελευταία ανάλυση, το ελεκτικό συνέδριο έδωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σε 9% του προπολογισμού, πράγμα το οποίο έχει γίνει και τα τελευταία πέντε χρόνια. Και για τους υπόλοιπους τομείς, για το 43% δηλαδή, η γνώμη εδώ πέρα είναι με, με επιφύλαξη και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί, ιδίως όταν απευθυνόμαστε στον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει δώσει αρνητική γνώμη για ένα 43% του προπολογισμού. Πώς θα τους εξηγήσουμε ότι τα χρήματά τους χρησιμοποιούνται όντως με εντιμότητα. Πώς θα μιλήσουμε για αποτελεσματικότητα όταν δεν προσπαθούμε καν να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα αυτή όσον αφορά την ε, σωστή ε, δαπάνη των πόρων. Θα ήθελα να απευθύνω προς το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο ένα ερώτημα. Θεωρούν ότι είναι σωστό να συνεχίσουν να εγκρίνουν προχρηματοδο... προχρηματοδοτήσεις σε τομείς όπου παρουσιάζονται πολύ μεγάλα σφάλματα όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία συνοχής κτλ και στο παρελθόν είχα υποβάλει ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αύξηση της προχρηματοδότησης και δυστυχώς δεν μου δόθηκε μία απάντηση για ποιο λόγο έχουμε αυτή την αύξηση στην προχρηματοδότηση και φοβάμαι ότι οι προχρηματοδοτήσεις τελικά ε, είναι γεμάτε σφάλματα. Έχουν να κάνουν τομεί που ε, παρουσιάζουν πολύ μεγάλα σφάλματα. Αναφερθήκατε σε τομεί που θα μπορούσαμε να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος. Δεν αφαιρθήκατε όμως σε βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επέλθουν στον προγραμματισμό του προπολογισμού στην καλύτερη σχεδίαση του προπολογισμού. Και κοιτώντας τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί και το ύψος των προχρηματοδοτήσεων, βλέπω ότι μας δίδεται εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μια πιο επαγγελματική και αυστηρή δουλειά κατάρτιση του προπολογισμού, σχεδιασμού του προπολογισμού, για να μην καταλήγουμε σε τόσο υψηλά ποσά προχρηματοδότηση ή σε τόσο υψηλά ποσοστά μη απορροφημένων κονδυλίων. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο και στη συνέχεια θα μιλήσει ο κύριος Καλντέιρα γιατί θα πρέπει συνέχεια να αποχωρήσει. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Καλδέιρα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και το σύνολο των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πολύτιμο αυτό έγγραφο το οποίο μας υποβάλλεται και για όλη την εργασία που έχετε κάνει με απόλυτη αυτονομία και ανεξαρτησία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υπηρεσίες του για την συνεχή βελτίωση που βλέπουμε από το ένα έτος στο άλλο στον αφορά την εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιες παρατηρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα με πέρυσι. Στα πλαίσια της αποστολής σας, στα πλαίσια της ανάλυσης που κάνετε, πέρα από τα λάθη, έχετε εντοπίσει και απάτη. Ξέρετε ότι κάνω εγώ μια πάρα πολύ σαφή διάκριση ανάμεσα στα σφάλματα, πολλές φορές στην απόφευκτα, και ανάμεσα στην απάτη, η οποία θα πρέπει να πεταχθεί, να καταπολεμηθεί. Δεύτερο τώρα ερώτημα, όσον αφορά του ιδίους σπόρους και όσον αφορά την ποιότητα του τελωνιακού μα συστήματος. Η Τελωνιακή Ένωση αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η εργασία γίνεται από τις εθνικές αρχές. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις νέες διευρύνσεις έχουν τροποποιηθεί. Επομένως, η ποιότητα της εργασίας που γίνεται από τις εθνικές αρμόδιες τελωνιακές αρχές μας επιτρέπουν να έχουμε μια σημαντική ανάκτηση όσον αφορά τους, ιδιουπο... τους ίδιους Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους δασμούς, γιατί ε, ένα 75% έρχεται στα κράτη-μέλη, ενώ 25% δίδεται από τους δασμούς αυτούς για τις διοικητικές δαπάνες και είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε για τη συλλογή των δασμών να μπορούν να συμβάλλουν για την καλύτερη κατάρτιση των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η έλλειψη απλούστευσης οδηγεί σε πάρα πολλά σφάλματα και λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η πολυπλοκότητα ορισμένων δραστηριοτήτων. Δεν έχω ακριβώς μπροστά μου τώρα το κείμενο, νομίζω ότι είναι στο σελίδα 31, τουλάχιστον στη γαλλική εκδοχή, εκδοχή. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ο νομοθέτης αυτός που ευθύνεται για την πολυπλοκότητα ορισμένων διαδικασιών. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε κάποιες διαδικασίες, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. διανύσαμε μία προεκλογική περίοδο για τις ευρωπαϊκές εκλογές ιδιαίτερα δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ προσεκτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνει τέτοιες δηλώσεις, γιατί πειράζει και αυτή πολύ τη γνώμη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τις διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ ότι ο νομοθέτης ή ο συνομοθέτης φέρει κάποια ευθύνη και δεν έχουμε όμως μόνο την πολυπλοκότητα ενός κανόνα, αλλά έχουμε και την εφαρμογή του κανόνα αυτού. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι προσεκτική κάθε φορά που κάνει τις δηλώσεις για το ποιος ευθύνεται για την πολυπλοκότητα ορισμένων νομοθετικών διατάξεων. Αναφερθήκατε επίση στην πολυπλοκότητα που έχει εντοπιστεί σε κάποιου τομεί όπω η έρευνα και σε άλλου τομεί. Όσον αφορά τα όργανα υψηλού βαθμού εποπτείας. Κύριε Καλτέρα, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο τα πορίσματα των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων καθώς επίσης και τα πορίσματα των ανώτατων οργάνων ελέγχου. Οι συνθήκε τη Λισαβόνα αλλά και οι προηγούμενε συνθήκε σα δίνουν τη δυνατότητα ω Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να ζητήσετε από τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια όλε τι απαραίτητε πληροφορίε και όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία χρειάζεστε για να επιτελέσετε το έργο σα. προτίθεστε εσείς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή που σας δίνεται προκειμένου ακόμα και στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου να χρησιμοποιήσετε κάποιες εθνικές πηγές. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο, πρέπει να σας πω ότι για την απαλλαγή του προπολογισμού 2007 έγινε μια πολύ σκληρή δουλειά και πολύ σκληρές θα έλεγα διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε ότι για το Συμβούλιο δεν υπάρχει κάποια γνωμοδότηση, ενώ για τα άλλα θεσμικά όργανα, π.χ. για την Επιτροπή των Περιφερειών, έχετε εκφέρει κάποια γνώμη. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την άποψη του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη λειτουργία του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρντέρα και τους 26 ε, συναδέφους του στο, σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο για την ε, έκθεση. Ίσως πολλά υπάρχουν και μπορούμε να τα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν άλλοι προλαλήσαντες. Μια συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω. Το ελεγκτικό συνέδριο κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και των ευρωπαϊκών πολιτικών, τι έχει κάνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, θα έλεγα. Μια, ένα σύνολο πληροφοριών που είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με τον προπολογισμό των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μα, για την επίτευξη των στόχων μα, για την αποκατάσταση εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν θα ήταν καλή ε, ιδέα στην ετήσια έκθεση να συμπεριληφθεί μια παράγραφο για την αποτελεσματικότητα και τι θετικέ επιδόσει των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Καλτέιρα θα λάβει τώρα τον λόγο παρακαλώ. Σα... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών για τα θετικά λόγια που έχουν πει για μένα και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Όντως όλοι συνέβαλαν στο να υποβληθεί σήμερα η ετήσια έκθεση σε εσά. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τα καλά ενθαρρυντικά σας λόγια. Σαφώς είμαστε εδώ πέρα για να εργαστούμε περισσότερο με τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων και συγκεκριμένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσά και στη συνεργασία που μπορεί να έχει το ελεκτικό συνέδριο με το δικό σας θεσμικό όργανο και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία αυτή στο μέλλον. Δεν θα είμαι σε θέση να απαντήσω σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ξεχωριστού τομεί πολιτική και να ομαδοποιήσω κατά κάποιον τρόπο τι ερωτήσει. Όσον αφορά τους λογαριασμού αυτού καθ' αυτού, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να εκτελέσει το έργο του προκειμένου να εξασφαλίσει λογικές και αποδεκτές εγγύσεις για τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ότι δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει να προβλέπονται λάθη, να μην υπάρχουν λάθη, ώστε να τον λιγότερα σφάλματα. Η φράση που χρησιμοποιούμε στη συνέχεια στο κείμενο, ότι ε, οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν ξεκάθαρα και δίκαια, αξιόπιστα, φέρλει τους ε, οικονομικούς, ε, την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά περιέχει την έννοια της αλήθειας των λογαριασμών αυτών. Όσον αφορά το εγχείρημα αυτό, να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, αποτελεσματικότητα και απλούστευση, εμείς δεν ζητάμε περισσότερα συστήματα. Δεν θέλουμε αύξηση και υπερβολικούς ελέγχους. Ήδη κάνουμε πολλούς ελέγχους. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι να το κάνετε, να το κάνετε με αποτελεσματικότητα. Γιατί κάθε φορά που τα συστήματα είναι αποτελεσματικά, τότε το επίπεδο των παράτυπων πληρωμών μειώνεται με την πάρδα του χρόνου. Σας δώσαμε και ένα παράδειγμα στα πλαίσια του τομέα γεωργίας. Αλλά ακόμα και στη Γεωργία, ακόμα και στο παρελθόν είχαμε παραδείγματα όπου υπήρχε περιθώριο για περαιτέρω απλούστευση. Στον τομέα της ανάπτυξης υπαίθρου, η πολλαπλή συμμόρφωση και τα περιβαλλοντικά μέτρα ήταν αντικείμενα πολιτικής όπου θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες απλουστεύσεις η απλούστευση ουσιαστικά σημαίνει μην περιπλέκετε τα πράγματα περισσότερο από ό,τι απαιτείτε. Δεν λέω ότι πρόκειται για περισσότερη ή λιγότερη γραφειοκρατία. Πρόκειται για μεγαλύτερη ξεκάθαρη ε, αντιμετώπιση των στόχων μας. Διαφάνεια και περνά στο ζήτημα αυτό της διαφάνειας. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει στα πλαίσια των συζητήσεων που κάνουμε για τον προπολογισμό. Και το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι νομοθέτης. Νομοθέτης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όταν είπατε λοιπόν ότι σας καλώ να τραγωνίσετε τον κύκλο, θα πρέπει καταρχάς να δείτε εσείς εδώ πέρα πώς είναι δυνατόν να γίνει πράξη όχι ο τετραγωνισμός του κύκλου, αλλά ο συνδυασμός αποτελεσματικότητας και απλούστευσης πιστεύω ότι είναι δυνατός. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο παρατυπιών αλλά ακόμα και απάτης που έχουμε δει στα πλαίσια των διατροτικών ταμείων. Διορθώνω, δεν πρόκειται για απάτη. Κύριε Οντή, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας και των ελέγχων που κάναμε, είδαμε ότι είχαμε δύο περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως περιπτώσεις απάτης, ενώ κάναμε πάρα πάρα πολλούς ελέγχους, περίπου 40 ή 45, για πάρα πολλές πληρωμές, τις οποίες είχαν εντοπιστεί απλώς παρατυπίες και έχουμε ενημερώσει προφανώς την Όλαφ για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Συνεργαζόμαστε, όπως ξέρετε, πολύ καλά με την Όλαφ. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό το 11% στο οποίο αναφέρθηκαν ορισμένοι ομιλητέ. Σας καλώ να δείτε τι λέμε στην παράγραφο 6 σημείο 6 στη σελίδα 124. Τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Λέμε ότι ο δικός μας έλεγχος έγινε σε ένα σύνολο 24,8 δισεκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τις ε, αποζημιώσεις. Αυτό εξετάσαμε εμείς στα πλαίσια της έκθεσής μας. Και αν πάτε στην ε, παράγραφο στην οποία αναφέρθηκε ο προλαλής σας 6.17 θα δείτε ότι υπάρχει μια μικρή υποσημείωση που λέει ότι το 11% θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στο ποσό των 24,8 εκατομμυρίων και όχι στα 46 δισεκατομμύρια που είναι το συνολικό ποσό για το 2008 για αυτόν τον τομέα. Όπως σας είπα, εξετάσαμε τις πληρωμές για την περίοδο 2000-2006 και ένα πολύ σημαντικό τμήμα ήταν προκαταβολή για την περίοδο 2007-2013 και οι προκαταβολές είναι πολύ σημαντικές και τίθεται το ζήτημα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι προκαταβολές ή όχι. Δεν είναι αρμόδιο όμως το λεκτικό συνέδριο για να πάρει μια τέτοια απόφαση. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αποφασίσει να αυξήσουν τις προκαταβολές εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης. Αν διαβάσετε το κεφάλαιο 3 σημείο 2 θα δείτε ότι κάνουμε κάποια αναφορά στα ποσά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε αν τα ποσά αυτά που αποτελούν προχρηματοδότηση και προκαταβολή έχουν απορροφηθεί σωστά, έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στον κύριο Οντί για αυτό που είπε για τη συνεργασία με, τη, με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και του, τους εθνικούς οργανισμούς, τα εθνικά όργανα ελέγχου. Σαφώς θέλουμε να αυξήσουμε την συνεργασία αυτή και θέλουμε να γνωρίζουμε πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανά... Ανάκαμψης και τους πόρους προβλέπω. Και θέλουμε όμως να δούμε επίσης και ποιοι είναι οι άλλοι τομείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους ιδίους πόρους της Ένωσης. Το Δεκέμβριο θα συζητήσουμε πώς θα αυξήσουμε καλύτερα και πώς θα βελτιώσουμε τη συνεργασία με τα νότα όργανα ελέγχου, τα εθνικά και με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Μπορώ επίση γραπτό να απαντήσω σε οποιασδήποτε άλλε ερωτήσει δεν είχα το χρόνο να καλύψω αυτή τη στιγμή. Και θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχή να έρθω οποτεδήποτε εσεί, κύριε Πρόεδρε, τα μέλη τη Επιτροπή στο Κρίντα Αναγκαίο, πάλι εδώ στην Επιτροπή σα για να απαντήσω σε άλλε ερωτήσει, είτε εγώ είτε μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όσον αφορά το αν θα πρέπει να κατανομαστούν κάποια κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των εθνικών συνοπτικών εκθέσεων, που έχουν ως στόχο να παρέχουν όλες αυτές τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτές οι εκθέσεις επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζει ποιες είναι οι επιδόσεις του κάθε κράτους μέλους και οι εκθέσεις αυτές επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να δει πώς εφαρμόζεται η συγχρηματοδότηση, πώς εφαρμόζονται οι προσαρμογές του προπολογισμού. Εμείς δεν έχουμε ως στόχο να ε, δούμε πώς ακριβώς συμπεριφέρεται κάθε κράτος μέλος. Καθήκον μας βάσει τη συνθήκη είναι να μιλήσουμε για την συνολική εκτέλεση του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό κάνουμε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση ανάμεσα στο, στην εξέταση του κοινοτικού επίπεδου και τη χρήση που γίνεται έπειτα από τα κράτη-μέλη. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ένα 80% των πόρων τυχαίνει διαχείρισης ε, από τα κράτη-μέλη. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να πω ότι με την αθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού με τις νέες εξελίξεις όσον αφορά την κατάρτιση του προπολογισμού και με την αναθεώρηση των νέων δημοσιονομικών προοπτικών μετά το 2014 έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία για να προχωρήσουμε περισσότερο με την απλούστευση, για να σχεδιάσουμε καλύτερα τους στόχους πολιτικής, για να επιφέρουμε την προστιθέμενη αξία των ε, πόρων και των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Eh, θα συνεχιστεί τώρα η συζήτηση. Ο κύριος Κάλλας θα πάρει το λόγο σε λίγο. Ο κύριος Γκάια μου ζήτησε πρώτα το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, συμπίπτει πολύ καλά αυτό, διότι η παρατήρηση που ήθελα να κάνω δεν στρέφεται τόσο πολύ στον κύριο Καλντέρα και τα άλλα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά περισσότερο δύο παρατηρήσεις ήθελα να κάνω και μία επερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρατήρηση είναι για τις προπληρωμές. Δεν ήμουν ακόμα στην Ευρωβουλή τότε, αλλά από τους συναδέλφους μου κατέστησε σαφές ότι αυτό το σύστημα προπληρωμών ήταν κάτι το οποίο θελήθηκε ως αντίδραση στην οικονομική κρίση σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πολύ γοργά να διατίθεται χρήμα σε αυτά ώστε τα προγράμματα αναδιάρθρωσης να μπορούν να λειτουργήσουν όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που ελπίζουμε εμείς ότι μέσω των ταμείων συνοχής και των, του Ταμείου Συνοχής και των κονδυλίων του θα εδρεωθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε, τα κονδύλια αυτά θα πρέπει προς κάθε κατεύθυνση να δαπανώνται και να μην έχουν αποτέλεσμα. Το αντίθετο, τα μέτρα τα οποία μέσω προπληρωμών στα κράτη-μέλη διατίθενται ήταν κάτι το οποίο θελήσαμε εσκεμμένα ένα ως μέτρο για να καταπολεμηθεί η οικονομική κρίση. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και να το θυμόμαστε και είναι και σημαντικό αυτό όταν ενδεχόμενα κατά τη διάρκεια του απογεύματος με εκπροσώπους του τύπου θα συνέλθουμε από κοινού για να δούμε αυτά τα πράγματα. Και εδώ να μην υπάρξει κάποια άλλη παρέκκληση στη συζήτηση από αυτή την τοποθέτηση και από τις προπληρωμές προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε θέμα λευκής επιταγής. Τώρα το επόμενο. Το άλλο είναι κάτι που για άλλη μια φορά ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό και που στη συζήτηση μάλλον θα είναι ένα χρήσιμο σημείο και αυτό. Για τα διαθετικά ταμεία έχουμε μία αλλαγή όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία και διατάξεις με τη νέα περίοδο στήριξης από το 2008 και θα πρέπει για άλλη μια φορά, το πω να, να προσέξουμε ιδιαίτερα, περισσότερο να προσέξουμε στην, ας το πω διασφάλιση ή αντιμετώπιση των περιπτώσεων του Ταμείου Συνοχής ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις με τις ε, διατάξεις ε, εκτέλεσης. Αυτό θα ήταν, να το πω έτσι, θα αφορούσε κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να υπογραμμίσουμε την χρησιμότητα αυτών των μέτρων. Τελευταίο θέμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνεργάτες μου, α, τυχαία μάλλον, σε σχέση με ένα αίτημα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους εμπλεκόμενους το ανακάλυψαν για μια διαδικασία απλούστευσης όσον αφορά τις ε, αιτήσει και τα έντυπα. Όλοι εκείνοι με τους οποίους ε, είχαν έρθει σε επαφή μαζί μου και συζήτησαν αυτά τα θέματα μαζί μου έλαβαν την ειδοποίηση να υποβάλουν προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Δεκέμβριο προτάσεις τους για βελτίωση της, των, των ε, όρων του παιχνιδιού. Επανειλημμένα είδα και το πρόσεξα ότι από εκείνους τους ε, που από πλευράς κάλυψης ε, καλύπτονται για παράδειγμα στο Μητρό Λομπίστων δεν έχουν ενημερωθεί για αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Θα με ενδιαφέρε να μάθω ποιος είναι ο λόγος για αυτή την κατάσταση, σε τι οφείλεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν αρκετά τα αιτήματα τα οποία ε, υπευλήθησαν αρκετές προτάσεις και προς το ελεγκτικό συνέδριο έγιναν παρατηρήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κύριο Κάλλας. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κάλλας, διότι κάτι πτυχέ, κάποιες πτυχές αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων και το θέμα που αφορούν, αφορά και τις παρατηρήσεις Χατζημαρκάκη και ε, Λιμπεράτσκι. Κατά πόσον είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή εδώ σε θέση να αντιμετωπίζει να αντιτίθεται σε εισαγωγικά έναντι των κρατών μελών, να, αντιμετωπίζει τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε για να διασφαλιστεί διαφάνεια και κυρίως αυτό θα σημαίνει πρώτα και κύρια ότι αυτό θα πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των πολιτών όσον αφορά τις ε, εκτελέσεις των πληρωμών. Και ο κύριος Γκάιερ έθεσε θέματα, ο κύριος Κάλλας έχει τον λόγο λοιπόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ πολύ εσάς Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια που απευθύνατε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τούτου λεφθέντας αρκετά σημαντικά θέματα έχουμε εδώ. Πρώτον έχουμε το θέμα για τα κράτη-μέλη και το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα στη διαχείριση των πραγμάτων με τα κράτη-μέλη. Πρώτα και κύρια θα ήθελα να πω ότι και πάλι εδώ για την έκθεσή μας που παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Το να κατονομάζουμε λοιπόν κράτη-μέλη είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Δεν ήταν πραγματικότητα πριν από πέντε χρόνια. Πολύ σπάνια αναφερόντουσαν ονομαστικά κράτη-μέλη τότε από πλευρά μα. Δεύτερο στοιχείο. Και το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό από πλευρά του επεσήμανε και στοχοθέτησε με ότι μεγάλο μέρος των σφαλμάτων που ανείχνευσε στην Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο ή Αγγλία περισσότερο για να είμαι ακριβέστερος αυτός ο, το να κατονομάζουμε και να καταγγέλουμε είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε και θα συνεχιστεί ως προσπάθεια σίγουρα σε συγκεκριμένες πτυχές για την αλλαγή ας το πω έτσι της κουλτούρας ε, του κλίματος είναι ε, ε, εντυπωσιακό. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μεγάλη αντίσταση να αναφέρονται κράτη-μέλη σε οποιοδήποτε έγγραφο, ακόμα και σε έγγραφα του ελεγκτικού συνεδρίου. Σήμερα ονομάζουμε, ονοματίζουμε όμω κράτη-μέλη και καταγγέλουμε πράγματα. Πώ μπορούμε να καταλήξουμε στην κοινή αυτή διαχείριση, στα ετήσια στοιχεία, στι επισκοπήσει και να βελτιωθούν τα πράγματα. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί και το νομικό πλαίσιο και η νομική βάση. Ξέρετε ότι οι αιτήσιε αυτέ συνόψει βασίζονται σε συνδιοργανική συμφωνία. Χρειαζόμαστε όμως τελικά κάτι και στο δημοσιονομικό κανονισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ καταλήγω στη μεγάλη ευκαιρία που αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο Καλντέιρα. Κατά το τέλος των, τε, παρατηρήσεών του ακροτελεύτιων παρατηρήσεων για τη συζήτηση για δημοσιονομικές πτυχές που θα ξεκινήσει και επίσημα εντός ολίγου. Συνοδεύεται από δημοσιονομικούς κανονισμούς και διατάξεις και θα πρέπει εκεί να προβληματιστούμε και να δούμε τις εξελίξεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με προτάσεις, προτάσεις της Ευρωβουλής και προτάσεις του Συμβουλίου για την τελική απόφαση που θα ληφθεί. Πρέπει να αντανακλά τις πραγματικότητες και τα προβλήματα αυτό. Και αυτό είναι μια από τις μεγάλες ευκαιρίες για την απλούστευση. Αναφέρθηκε ότι περίπλοκοι κανόνες, πολύπλοκα πράγματα και άλλα σε άλλα οφείλεται αυτή η κατάσταση και ο κύριος Καλντέιρα πάλι από πλευράς του και μπορώ να τον αναφέρω σε παράθεμα όταν λέει ότι έχει και όρια η απλούστευση έχει και όρια στα οποία φτάνει πια α, ως εγχείρημα αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες όπου και με ενθουσιώδη τρόπο από πλευρά του πολλέ φορέ κάποιοι υπάλληλοι περιπλέκουν τα πράγματα στον υπερβάλλοντα ζήλο του. Όμως το κύριο θέμα από το 2002-2006 είχαμε 545 προγράμματα στα διαφορετικά ταμεία. 545 προγράμματα. Λοιπόν, κάθε πρόγραμμα έχει και τη δική του ξεχωριστή νομική βάση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκινούν όχι από αυτήν εδώ την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όλα αυτά έχουν τα, τις ρίζες τους ε, στη δική μας ε, διεύθυνση, στις δικές μας διευθύνσεις χάραξης πολιτικής, κατάθεσης πολιτικής, πάνε μετά στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και μετά και στο Συμβούλιο σε σχέση με την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο. Το να σχεδιαστούν και να κατατιστούν τώρα νέε δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να περιορίσουμε κάποια προγράμματα και να περιορίσουμε το εύρος όλων αυτών. Τώρα, για τα νέα προγράμματα και για το αν θα είναι απλούστερα, για την Γεωργία για παράδειγμα. Η Γεωργία έκανε πολλές προσπάθειες για να βελτιωθούν ε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και πέτυχαν σχεδόν ε, καθαρά ή πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με την παραδοσιακή χρηματοδότηση της Γεωργίας Όμω το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη τη υπαίθρου. Και τώρα τίθεται το ζήτημα, το ερώτημα, πώ μπορούμε να πετύχουμε του στόχου, να συγκεράσουμε του στόχου. Και αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο Καλντέρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από άλλου ευρωβουλευτέ και αυτό. Α, λοιπόν, τούτων λεχθέντων, αν χώρε αν κράτη-μέλη που είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί ε, που πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. αλλά κάποιοι που πληρώνουν και κάθε χώρα πληρώνει το μερίδιό τη ούτω ή άλλω στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αν ρωτήσουν αυτοί πού πάνε λοιπόν αυτά τα χρήματα, λέω εγώ α αναφέρουμε συνολικά ποσά ανακράτη-μέλη ή αναπεριφέρειε ή ουσδήποτε άλλου τομεί και μετά ρωτάνε πού, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα τίθενται ερωτήσεις. Πρέπει να περιγραφούν λοιπόν κάποιοι στόχοι και καμιά φορά είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και από πλευρά ενό και, και ιδίου προγράμματος για να καθορίζονται αυτά θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία, να υπάρχει αξιολόγηση και έλεγχος ταυτόχρονα. Η κύρια πρότασή μου φυσικά είναι ότι σίγουρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην Επιτροπή για να μειωθεί ο αριθμός των προγραμμάτων και το εύρος τους και να απλουστευτεί το εύρο των πλαισίων ε, διατάξεων και κανονισμών. Όμως μια πολιτική θα παραμείνει που θα χαράζεται και θα καταρτίζεται. Και για τα κονδύλια των ε, δράσεων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που διατίθενται σε διάφορες δράσεις και όσον αφορά και επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις ε, πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους και πάλι θα ρωτήσουν οι φορολογούμενοι τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια, ακόμα και αν είναι απλούστεροι οι κανόνες. Και πάλι όταν θα υπάρχει κάποιο ποσοστό σφάλματος για κάποια περιφέρεια στην οποία θα δίνεται ένα ποσό, πάλι πρέπει να δούμε τι θα αναζητώνται ευθύνε. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι τα κράτη-μέλη αρχίζουν να κοιτάζουν πολύ προσεκτικά και το κόστος του ελέγχου που είναι μια σημαντική παράμετρος επειδή ενισχύουμε τις απαιτήσεις για ελέγχους και τώρα έχουν τα κράτη-μέλη ξεκινήσει να ανακαλύπτουν ότι σε κάποιους τομείς πρέπει να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να ε, έχουν καλή αξιολόγηση και να βαίνουν καλό τα πράγματα και να πιστοποιούνται ότι βαίνουν καλώς. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα σε σχέση με τα όσα ήθελα να πω. Και όλα αυτά σε σχέση με τα κράτη-μέλη όπως σαφώς υπογραμμίστηκε, βασίστηκαν σε πολύ καλή συνεργασία και στο συσχετισμό τη Ευρωβουλή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα και να δώσουμε συνέχεια σε αυτέ τι προτάσει. Αλλά να ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση η δημοσιονομική και για τι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ και την παρακολούθηση και συνόδευση των ε, μελλοντικών προτάσεων για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά την προπληρωμή, τι προπληρωμέ ε, που ε, πολλέ φορέ αναφέρθηκαν και με προπληρωμέ πάντα υπάρχουν υπάρχουν και ενέχονται κίνδυνοι. Και είναι σαφές αυτό. Και αν γενναιόδωρα προπληρώνονται με πληρωμές κάποια προγράμματα, πρέπει να είναι κανείς βέβαιος ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι στη συνέχεια. Γιατί μετά τίθενται τα θέματα ανάκτησης κονδυλίων αν κάτι δεν πάει καλά. Και όλα αυτά θεωρούμε εμεί ότι είναι απόλυτα νόμιμα σήμερα. Και όλα αυτά συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ε, ε, διάνοιξη μιας νέας διαχειριστικής περίοδου και την απουσία συγκεκριμένων καθυστερήσεων όσον αφορά στη συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη που πολλές φορές κρατούσαν χρήματα και δεν, συγχρη... δεν συγχρηματοδοτούσαν για να προχωρήσουν τα προγράμματα. Έχει προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις περιφέρειες και χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με συγκεκριμένες περιφέρειες για να διατίθενται κονδύλια έγκαιρα. Εμείς δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα και προσκόμματα. Δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα ε, αναχαιτήσουν την χρηματοδότηση αν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτό δεν θα σημαίνει όμως ότι οι κανονισμοί και οι κανόνες έχουν αλλάξει ή ότι οι απαιτήσει για τη χρηστή διαχείριση θα συρρυκνωθούν και θα μειωθούν. Καθόλου δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά βέβαια οι προπληρωμές είναι, οι προκαταβολές είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Με αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω με άλλα λόγια εδώ και σήμερα και πάλι υπογραμμίζοντας ότι σήμερα έχουμε την, είχαμε την παρουσίαση της έκθεσης των εκθέσεων του, του ελεγκτικού συνεδρίου εμείς έχουμε ξεκινήσει όμως ε, ε, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα συζητώντας ε, τα θέματα των εκθέσεων από πλευρά μας όλοι οι επίτροποι με ιδιαίτερη χαρά και προθυμία προσέρχονται για να λογοδοτήσουν και να σας ενημερώσουν εδώ δεν μπορώ να ε, προκαταλάβω τίποτα. Είναι η δουλειά μας βέβαια αυτή ως επίτροπο να κάνουμε τη δουλειά μας με πλήρη συνέστηση ευθυνών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις ε, και από ό,τι βλέπω όχι. Α, ο κύριος Σοντή, παρακαλώ. Σύντομα. Πρόεδρε, ξέχασα να πω πριν από λίγο στον Πρόεδρο Καλτέρα ότι πάντοτε δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς γίνεται η έκθεση του, του συνεδρίου που έχει ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου να μην ανακοινώνεται, κοινοποιείται σε εμά παρά σήμερα. 10 Νοεμβρίου. Εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε τη στιγμή που υπογράφεται η έκθεση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Γιατί όλοι κάθονται και περιμένουν την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου χειρότερα από ότι τα απομνημονέματα του Ζακ Σιράκ στη Γαλλία έχει καταντήσει. Άπρεπε λοιπόν να μπορούμε να τα έχουμε τη στιγμή που υπογράφονται. Και συνάδελφε Οντί, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όπως γνωρίζετε έγινε μια διαπραγμάτευση με το συνέδριο και το συνέδριο ε, θεωρεί πως είναι πιο σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο την, έχει κατά κάποιο τρόπο την αποκλειστικότητα με τον τύπο. Το γεγονός ότι εμείς το πήραμε τα τελευταία στιγμή ε, σχετίζεται με το γεγονός ότι το συνέδριο που θεωρεί αυτό την εργασία την πιο σημαντική ολόκληρο της χρονιάς να παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο κατευθείαν προς τον τύπο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας για το γεγονός ότι και το έχουμε ήδη πει και άλλες φορές, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να ε, μπορούμε να κάνουμε μια ευρύτατη συζήτηση χωρίς να έχουμε μετρημένα τα λεπτά γιατί πρέπει να πάει να κάνει ανακοίνωση τύπου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε και να το πετύχουμε, να τα έχουμε την έκθεση τουλάχιστον λίγες μέρες νωρίτερα. Μια παρατήρηση. Εγώ έχω κάνει έλεγχο στο παρελθόν. Εγώ ποτέ δεν έχω δει κάποιον ελεγκτή να κάνει συνεντεύξεις τύπου. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το να κάνει ένας ελεγκτής ε, ε, συνεντεύξεις τύπου. Συμφωνώ. Όλοι συμφωνούν από ό,τι βλέπω. Εμείς δεν πάμε λοιπόν στην συνέντευξη τύπου, πάμε για δουλειά και θα τα ξαναπούμε στις 2 Δεκεμβρίου.